colleagues, please. Σας παρακαλώ, είναι 9 και 10. Ας ξεκινήσουμε. Good morning to everybody. Καλημέρα σε όλους σας. Το πρώτο σημείο είναι οι αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν χθες στο τέλος της συνεδριάσεως όσον αφορά τη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπαν οι υπάλληλοι τι γίνεται, οι υπάλληλοι παρακολουθούν τις εργασίες και καταλήξαμε δέσμευση όλων των συντονιστών της Επιτροπής μας να υποστηρίξουμε τις εργασίες που γίνονται ούτως ώστε να γίνει ταχύτερο δυνατόν ε, ετοιμαστεί αυτή η δικτυακή πύλη, το ταχύτερο δυνατόν ε, για να μπορέσουμε τελικά να καταβάλουμε προσπάθειες και ξεπεράσουμε τις Όσον αφορά τις διάφορες αποστολέ, τι ερευνητικέ για το 2013, οι συντονιστέ συμφώνησαν ότι πρέπει να διοργανωθούν αποστολές η πρώτη να στην Ισπανία, στην περιοχή της Γαλλικίας και η δεύτερη στην Ελλάδα. Μετά επιφυλάχθηκαμε για αποφάσεις ενδεχόμενες άλλες αποστολές για το 2013 και θα το συζητήσουμε σε μια περαιτέρω συνεδρίαση ε, στα πλαίσια των κατεπηγουσών αναγκών που θα δημιουργηθούν από διάφορες αναφορές θα υποβληθούν στα μέλη της Επίτροπης. Αποφασίστηκαν και οι δύο ακροάσεις. Η πρώτη ήδη που ανακοινώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια που θα πραγματοποιηθεί μαζί με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών που θα πρέπει να λάβει χώρα στις 19 Φεβρουαρίου του 2013 η δεύτερη όμως, για την οποία είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη σύνοδο για να δημιουργηθεί η Φορολογική Ένωση, ξεκινώντας από την αναφορά που υποβλήθηκε από συναδάλφους Νταφ και Λάινεν. Αυτή η δεύτερη ακρόαση ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Είμαστε σε μια φάση αρχική όσον αφορά τις συστάσεις που παρουσίασαν οι συνάδελφοι βουλευτές, όσον αφορά τη, τη, κάποιες αναφορές και την αξιολόγηση της γραμματείας, έγινε αποδεκτή η πρόταση του κ. να επανεξεταστεί η σύσταση που αφορούσε την αναφορά 540 του 2012, οι άλλες αιτήσει του κυρίου, τα άλλα αιτήματα του κυρίου Ντουρκάης αποσύρθηκαν και οι συστάσεις του κυρίου Μπουλάντ ε, ανεβλήθησαν για συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Όσον αφορά το σημείο 4, που αφορούσε την πρόταση της ομάδας του ΕΛΚ για έναν ορισμό του κανονισμού για την διοργάνωση των αποστολών της Επιτροπής Αναφοράς και όσον αφορά την εφαρμογή του 202, αποφασίστηκε να αναβληθεί η συζήτηση εν αναμονή αναλόγων προτάσεων από πλευράς των άλλων ομάδων που παρίστανται στην Επιτροπή. Το αίτημα του κυρίου David Skinner, που είναι στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας των συντονιστών, να υποστηριχθεί δηλαδή η δική του αναφορά με ένα αίτημα ψηφίσματος στην Ολομέλεια, είναι ένα αίτημα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τα μέλη, από τους συντονιστές, διότι τι μεταξύ άλλων μεταξύ των άλλων αντιρρήσεων που εξέφρασαν οι συνάδελφοι υπήρξε και η εκκρεμωδικία κάποιων υποθέσεων που θα δημιουργούσε κάποια σύγκρουση με τις δικές μας δραστηριότητε, οπότε αποφασίστηκε να μην υποβληθεί το ψήφισμα για το θέμα που υποστηρίζει ο κύριος Σκίνερ εγκρίθηκε το σχέδιο, το προσχέδιο μερίσιας διάταξης για την επόμενη σύνοδο της 6ης ε, Νοεμβρίου, το οποίο σχέδιο μερίσιας διάταξης δυναμίτησε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τον κατάλογο των αμφισβητουμένων ε, αναφορών που προβλήθηκαν και όσον αφορά των questionable submissions, όσον αφορά τις αποστολές που ε, είχαν προγραμματιστεί για το τέλος Οκτωβρίου, η αποστολή στην Πολωνία δυστυχώς ε, ακυρώθηκε διότι τα μέλη των ομάδων απέσυραν το ενδιαφέρον τους και τη διαθεσιμότητά τους και η αντιπροσωπεία βρέθηκε χωρίς μέλη ε, ε, με την εξαίρεση του συναδέλφου Τέιλορ που επιβεβαίωσε ότι είναι διαθέσιμος αλλά αποφασίστηκε μετά από όλα αυτά να αναβληθεί και αυτή η αποστολή για τον επόμενο χρόνο, για το 2013 θα ξαναπροταθεί το 2013. Όσον αφορά την ε, αποστολή στην Ιταλία, έγινε μια συζήτηση όσον αφορά τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος των συντονιστών που υπευλήθη στην προηγούμενη συνεδρίαση όσον αφορά την ερμηνεία των, του κανονισμού, όσον αφορά το διορισμό, αν ο πρόεδρος τη Επιτροπή μπορεί να ηγηθεί τη αντιπροσωπεία όταν η αντιπροσωπεία πάει στη χώρα στην οποία εκλέγεται ο, ο, πρόεδρος. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, τη γνωμοδότηση εξεφράστηκαν αντίθετε απόψει όσον αφορά την πρόταση για το ποιο θα είναι πρόεδρος της ε, αποστολή, Η S&D, η GUE, η Πράσινη και άλλοι ήταν αντίθετοι όσον αφορά η πρόεδρο να είναι επικεφαλή τη αντιπροσωπείας, οπότε η πρόταση απερίφθη από την ε, πλειοψηφία των συντονιστών και αποφασίστηκε το θέμα αυτό να διαβιβαστεί στη διάσκεψη των Προέδρων ούτως ώστε να αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων επί του θέματος εμπιστοσύνη δυνάμει του άρθρου 19 του Στερικού Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Δύο πράγματα. Να πω καταρχάς στου αδέλφου εδώ ότι δεν είμαστε κατά της Πρόεδρο. Αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε. Το μόνο που ψηφίσαμε ήταν ότι πρέπει να τηρηθούν οι παλιοί κανόνε ότι δηλαδή μέλος ε, υπήκοος τη χώρα δεν μπορεί να είναι επίσημα μέλο μια αντιπροσωπείας που επισκέπτεται τη χώρα του. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ή την πρόεδρο της Επιτροπής. Ό,τι αφορά τώρα την γνωμοδότηση της νομικής ε, υπηρεσίας, είναι σαφές ότι έχουμε κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίσουμε για τη σύνθεση των αντιπροσωπιών. Δεν είναι παράνομο και νομίζω ότι αυτό ήταν ξεκάθαρο. Έχουμε όμω το κυρίαρχο δικαίωμα. Και επαναλαμβάνω, δεν στρεφόμαστε κατά τη Προέδρου μα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση. Επίση, σε ό,τι αφορά το αρχικό πρόγραμμα και τη σύνθεση τη προσωπίας θα ήθελα να επανέλθουμε για το ιταλικό ζήτημα και κάτι άλλο θέλω να αναφέρω. Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά μπερδεύτηκα που ετέθη αυτό το ζήτημα για την όκρα. Είχα δει ότι εκτός της φωτογραφίας προέκυψαν και νέες πληροφορίες. Αυτό είχε προκύψει ήδη όταν είχα ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή η εν λόγω αναφορά. Θέλω να γραφεί λοιπόν στα πρακτικά. Όχι να το συζητήσουμε τώρα, απλά να ζητήσω να υπάρχει δυνατότητα όταν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, γιατί με εξέπληξε ε, ξέρω ότι ήταν σε σημείο του πρόεδρου, αλλά κάποιος μπορεί να το ζητήσει να μην είναι έτοιμο. Πράγματι όμως υπήρχαν νέες πληροφορίες. Και όχι μόνο φωτογραφία όπως υπόθηκε χθε, αυτό θα σας πω προς ενημέρωση. Προς ενημέρωση. Και παραλαμβάνω να επανέλθουμε στην αρχική εκδοχή του προγράμματος και της ε, σύνθεσης αντιπροσωπείας για την Άπολη και για τη Ρώμη. Ευχαριστώ. Κυρία Άουκεν, όπως γνωρίζετε για όλες τις αναφορές, ε, προστίθενται νέες πληροφορίες που αξιολογούνται θετικά από τα μέλη της Επιτροπής. Μπορούμε πάντα να ξανανοίξουμε το θέμα. Από τη στιγμή που θα δοθούν αυτά τα στοιχεία, οι συντονιστές μπορούν ε, να το συζητήσουν. Όσον αφορά την ε, αντιπροσωπεία για την αποστολή στην Ιταλία, δεν υπάρχει προηγούμενο σχήμα Οπότε είναι σαφές ότι το αίτημά σα, δεν είναι κατανοητό και μη παραδεκτό. Ο κύριος Ιτουργκάης έχει το λόγο. Eh. Δεν υπάρχει ένα θέμα, το είπατε, γιατί Νόρκα το συζητήσαμε στους συντονιστές σήμερα. Ίσως πρέπει να καταλάβουμε ότι γίνεται μόνο ανακοίνωση της Προέδρου για τα θέματα αυτά. Μάργαρετ, δεν ε, ξεκινάμε τη συζήτηση εκ νέου. Ε, θες να ξανασυζητήσουμε για αυτό το θέμα, μπορούμε. Χθε όμως ελήφθη η απόφαση για την όρκα και έχει ήδη κλείσει η εν λόγω αναφορά, γιατί έτσι αποφασίσαμε οι περισσότεροι από τους συντονιστές. Θέλετε να ψηφίσουμε, τι να σας πω, ή να λάβουμε μια άλλη απόφαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αποστολή στην Ιταλία, όπως και η Πρόεδρος και εγώ, ε, συμφωνώ το θέμα να παραπευθεί στη διάσκεψη των Προέδρων. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους να μην ξαναρχίζουμε να συζητάμε θέματα που τα συζητήσαμε και εφόσον ε, όταν υπάρχουν κάποια θέματα ανοιχτά πρέπει να τα συζητάμε όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων Θέλω οπωσδήποτε να το σημειώσω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη. Η αποστολή αυτή fact-finding στην Ιταλία θα ήθελα να παρακαλέσω να λάβετε υπόψη ότι χθε σίγουρα από πλευράς ε, επιχειρημάτων ε, δεν ήταν ε, η πιο αντικειμενική συζήτηση. Θα ήθελα παρακαλώ να ξανασυζητήσουμε, να, ξανα, να επιστρέψουμε στο θέμα επί της ουσίας του. Είναι δύσκολο να συζητήσουμε την ουσία για μας, για το ΕΛΚ. Είναι δυνατόν η πρόεδρος να είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας αλλά προς όφελος ε, των αναφερόντων παρακαλώ να καταλήξουμε ομόφωνα για τη σύνθεση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την επίσκεψη. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους συντονιστές και θα συνεχίσουμε τις επαφές από αυτού. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Καλώς. Αυτές είναι οι ανακοινώσει που είχα όσον αφορά τη συνεδρίαση των συντονιστών που έγινε χθε το βράδυ, που θα καταγραφούν στα πρακτικά μαζί με τις απόψεις εξέφρασαν αυτή τη στιγμή συνάδελφοι. Κλείνουμε λοιπόν το σημείο 11. Πάω στο σημείο 12 τη ημερησία διάταξη. Έχουμε την αναφορά 1550 του 2010 που υπευλήθη από πολίτη Μαλτέζικης Ιθαγένεια, που καταγγέλει ισχυρισμού περί ζημίας και απειλής για την ανθρώπινη υγεία από τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στα ναυπηγεία Παλούμπο στη Μάλτα. Δεν είναι παρούσα ή αναφέρουσα, οπότε για αυτή την αναφορά θα δώσω το λόγο αμέσως στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μάρκο Παδιώτη. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Όσον αφορά την αναφορά 1550-2010, δύο θέματα είχαν τεθεί. Πρώτο, ο θόρυβος δίπλα στα ναυπηγεία. Για το θέμα αυτό είπαμε ότι είχε υπάρξει διαδικασία λόγω έλλειψης ε, πρωτοβουλειών από πλευράς των ε, αρχών της Μάλτας, οι οποίες δεν είχαν καταλάβει το πρόβλημα. Η Επιτροπή απέσαιρε τη διαδικασία όταν μας έστειλαν τους χάρτες στο Ρίβου οι μαλτέζικες αρχές. Όσον αφορά την ε, ποιότητα του αέρα, έγινε μία μελέτη και οι αρχές της Μάλτας μας απήντησαν ότι δεν εφαρμόζεται η σχετική οδηγία επιτόπου, η PPC. Μετά υπήρξαν ε, επιστολές το 2011 και το 2012 μετά από επαφές της Επιτροπής με τις αρχές ε, της ε, Μάλτας και ζήτησε πληροφορίες για τη δραστηριότητα αυτού του ναυπηγείου και στις απαντήσεις τους οι αρχές που στις απαντήσεις 15 Ιουνίου 12 επιβεβαίωσαν ότι δεν υπόκειται στην οδηγία η εγκατάσταση αυτή και μόνο η οδηγία 1399 ε, είναι, ε, αφορά αυτή τη διαδικασία και μας είπαν ότι θα την ακολουθήσουν. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση. Δεν έχει υπάρξει νέο πιλωτικό πρόγραμμα, άρα παρακολουθούμε στενά την ε, κατάσταση μέσω διμερών επαφών. Η Επιτροπή και οι Εθνικές Αρχές θα συζητήσουν την κατάσταση για την αναφορά αυτή. Θα γίνουν περαιτέρω έρευνες και η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει μεθαύριο, 11 Οκτωβρίου. Οπότε δεν έχουμε περαιτέρω πληροφόρηση αυτή τη στιγμή, θα την έχουμε σε λίγες μέρες. Θα ζητήσουμε λοιπόν σε αυτή την συνάντηση ενημέρωση εάν έχει ε, εκδοθεί η τελική περιβαλλοντική έγκριση, ποιες είναι οι συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ε, μόνιση του αέρα και κατά πόσον εφαρμόζεται η οδηγία ε, για ε, τους διαλύτες. Εάν ακόμη δεν έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική άδεια, θα ρωτήσουμε γιατί. Ο Πίτερ Γιάν μου ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από πλευρά του συναδέλφου Μπούσουτιλ που θα ήθελε να είναι παρόν για τη συζήτηση αυτή τη αναφορά, αλλά δυστυχώ δεν είναι σε θέση να είναι εδώ. Τρει ερωτήσει θέλω να απευθύνω στην Κομισιόν που είναι σημαντικέ για αυτόν. Πρώτη, μπορεί να μα επιβεβαιώσει η Επιτροπή εάν οι οριακέ τιμέ το 2010 και 2011 σε σχέση με την ποιότητα του αέρα είναι συμβατέ με την ε, κοινοτική νομοθεσία. Δεύτερον, Μπορεί να μας επιβεβαιώσει η Κομισιόν εάν αυτά που ε, έχουν αναφερθεί για την ποιότητα του αέρα και του θορύβου είναι συμβατά με την νομοθεσία. Τρίτον, πότε θα μας δώσει οριστική απάντηση για το θέμα Παλούμπο η Κομισιόν. Από όσα μας είπατε, κατάλαβα ότι γίνονται διαπραγματεύσεις και συζητήσεις μεταξύ Επιτροπής Ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι μιλάς για τη 13, ε. Για τη 13, όχι για τη 12. Όχι, για τη 12. Για τη 12 λέει ο κύριος Γιάννη. Α, 12, ωραία. Σωστά, σωστά. Για τη 12 κύριε εκπρόσωπε της Επιτροπής. Για τη 12, για τη 12 βεβαίως. Βεβαίως αν κατάλαβα καλά, μας είπε η Επιτροπή ότι είναι σε επαφή με τις αρχές της Μάλτας. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε πότε θα λάβουμε την οριστική απάντηση και μέχρι τότε παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Πρώτη ερώτηση. Οι τιμές για το 10-11 και αν είναι εντός των ορίων και πάλι με συγχωρείτε, αλλά θα το συναντήσουμε μεθαύριο. Θα μας πούν τότε. Για το θόρυβο τώρα. Η οδηγία για τον ε, περιβαλλοντικό θόρυβο. Ζητούν από τα κράτη-μέλη πρώτα να υποβάλουν χάρτες θορύβου και μετά προγράμματα δράσης. Αλλά στην οδηγία γράφεται ότι ότι πρέπει να περιλαμβάνονται οι βιομηχανικοί χώροι που υπάγονται στην οδηγία EPPC. Επειδή μα είπαν οι αρχές της Μάλτας ότι για αυτή τη συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν ισχύει, δεν υπάγεται αυτή η εγκατάσταση στην οδηγία αυτή, άρα μπορεί να μην χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Οπότε δηλαδή ισχύουν οι εθνικές ρυθμίσεις για αυτή την εγκατάσταση. Τελευταία ερώτηση. Πότε θα κλείσουμε αυτή την αναφορά. Ενδεχομένω ε, μετά τις επόμενες συζητήσεις μας με την ε, Μάλτα. Ευχαριστώ. Πέτερ, μετά από αυτά που άκουσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει ακόμη κάποιες συνομιλίες με τις μαλτέζικες αρχές ε, συμφωνεί να μην είναι ανοιχτή αναφορά μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι επαφέ μετά να μα δώσουν οι πρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πληροφορία και να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία, τέλεια. Περνάμε λοιπόν στην υπαρχόν 13 αναφορά. Okay. Υπάρχει ένα πρόβλημα δεν, ναι, ήταν, δεν έχει έρθει ακόμη ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 13, οπότε περνάμε στην υπαρθμό 14, την αναφορά του Χωσέ Γκερέρο Δομή για Ισπανική Ιθαγένεια, εξ ονόματο τη πλατφόρμα Βεθινάλ προ το Τεραμνέτο, το VSA 33, σχετικά με την ηχορύπανση από αστικτικό αυτοκινητόδρομο στο κάτι τη Ισπανία, η οποία εικάζεται ότι παραβιάζει την οδηγία 2002 49 ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Παρίστατε ο αναφέρον, κύριε Γερέρο Δομήνγκες, καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτές. Ε, εκπροσωπώ την ε, ε, πλατφόρμα Βεθινάλ για τον αυτοκινητοδρομο c CE33, ο οποίος διέρχεται από το Κάντιφ της Ισπανίας. Πριν από 1,5 χρόνο εγγράφος ε, ζητήσαμε την παρέμβαση της Επιτροπής Αναφορών απέναντι στην Ισπανική κυβέρνηση με αναφορά μας. Τι συμβαίνει. Πριν από 20 χρόνια ε, κατασκευάστηκε μια παρακαμπτήρια οδός ε, για να παρακάμπτει λοφορία από τον τέταρτο αστικό αυτοκινητόδρομο που περνούσε ε, από το βορρά στο νότο και είχε δημιουργηθεί αυτός ο αυτοκινητόδρομος σε αστική περιοχή και διασχίζει και διαιρεί την πόλη το βόρειο κομμάτι της και επίσης το διαιρεί από το ανατολικό από το δυτικό παραγνωρίζει επίσης ε, κάποιους κανόνες που λέει ότι τέτοια αυτοκινητότητα, τέτοιες αρτηρίες θα πρέπει να απέχουν 100 μέτρα από κατοικίες, ενώ αυτή απέχει 5 με 10 μέτρα. Και κάθε μέρα πρέπει να είναι πάνω από 50.000 οχήματα. Λόγω τη μικρή απόσταση από τι κατοικίε και τι υψηλέ ταχύτητε που αναπτύσσουν τα οχήματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη χορύπανση στην περιοχή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται κυρίω ε, και στα κτίρια που είναι πολυόροφα. Ε, με βάση την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι επιπτώσεις από την έκθεση σε τόσο υψηλά επίπεδα θορύβου δημιουργεί κόφο, η έλλειψη ε, ικανότητα συγκέντρωσης, υπέρταση, αύξηση καρδιαγκιακών κινδύνων, ε, ε, διάφορες άλλες ευαισθησίες, ακόμη και απώλεια όραση μεταξύ άλλων και τα παιδιά που είναι τα πλέον ευάλωτα ε, μειώνονται και οι γνωστικές τους δυνατότητες. Ή, τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξη το 2008 στις, ε, περιοχές Γλωριέτα και Γράσια Σούσα Σαμποδέρ έχει δημιουργήσει κάποια ηχοπετάσματα, τα οποία ε, όμως δημιουργούν πρόβλημα ακόμη και λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ του αυτοκινητόδρομου και των κατοικιών, αλλά και γιατί υπάρχουν όροφοι που είναι πάνω από το ύψος των ηχοπετασμάτων αυτών. Υπάρχει λοιπόν η χορύπανση και μετά την τοποθέτηση αυτών των ηχοπετασμάτων και αυτό έχει αποδειχθεί με διάφορες μετρήσεις οι οποίες έγιναν από το προσωπικό του σχετικού εργαστηρίου της χάραξης αυτοκινητόδρων της ε, περιοχής των σχετικών αρχών από το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξη. Δηλαδή έχει επιβεβαιωθεί με μετρήσει ότι υπάρχει χορύπανση. Η έκθεση αυτού του εργαστηρίου λέει ότι οι επιτρεπόμενες τιμές θορύβου ε, ξεπερνούνται. Είναι υψηλότερα τα δεσιμπέλ. Ο επικεφαλής ε, το δικού δικτύου και επικεφαλής όμως του εργαστηρίου ε, διαφοροποιούνται και αναφέρονται σε ένα αυτοδιάταγμα του 96 της αυτόνομης περιφέρειας όπου ο θόρυβος που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, ο θόρυβος υποβάθρου λόγω της κυκλοφορίας ε, εξαιρούνται. Το περίεργο είναι ότι αυτό ο κανονισμό, αυτό το διάταγμα εδώ και νέα χρόνια είχε κυρωθεί αφού του τέθηκε σε ισχύ κρατικές ε, διατάξεις και τις αυτόνομες περιφέρειες σχετικά με την χορύπανση για να εφαρμόσουν στο Εθνικό Δίκαιο την Οδηγία 49 του 2002. Επομένως, ισχύει αυτή η οδηγία, αλλά και οι διατάξεις, ε, οι εθνικές και τις αυτόνομης περιφέρειας. Και φαίνεται ότι παραγνωρίζεται, και είναι ύποπτο αυτό, ε, παραγνωρίζεται ότι ένας από τους στόχους αυτής της οδηγίας και αυτών των διατάξεων είναι η μείωση του θορύβου από τις βασικές του πηγές, οι οδικές υποδομές και το τα περιλαμβάνονται σε αυτές τις ε, πηγές θορύβου. Μεταξύ τώρα των σχεδίων δράσης καταπολέμησης του θορύβου τη συγχωρήπας, τα οποία εκπονεί το Υπουργείο Ανάπτυξη για τη συγκεκριμένη περιοχή και ε, παραδόξω προβλέπεται η δημιουργία ανέγερση ηχοπετασμάτων. Αλλά περίεργο είναι ότι αυτό το μέτρο δεν έχει λύσει το πρόβλημα, γιατί το πόσο μάλλον το έχει επιδεινώσει. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν πρέπει να γίνουν πιο πολύπλοκες ε, παρεμβάσεις, όχι απλά να ανεγερθούν πετάσματα. Παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να αλλάξει χάραξη ε, να, είναι, ε, να βυθιστεί μέρος ε, της οδικής αυτής αρτηρίας. Και με αυτή την πρόταση, και εμείς είμαστε σύμφωνοι στην πλατφόρμα αυτή, αν δίπλα στα σπίτια μας έχουμε αυτό τον αυτοκινητό, τουλάχιστον να έχει βυθιστεί ένα κομμάτι του για να βελτιωθεί και η ποιότητα της δικής μας ζωής. Θα ήθελα να προβώ σε μια εκτίμηση. Πριν από έξι μήνες στείλαμε τους ισχυρισμούς μας ε, και τις απαντήσεις μας στην έκθεση της Κομισιόν. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Και ολοκληρώνω με το εξή. Ζητώ από την Επιτροπή σας να παρέμβει ώστε οι πολίτες οι οποίοι πλήγονται από αυτή την ε, επιβλαβή χορύπανση να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους τα οποία παραβιάζονται επανειλημμένως από τις αρχές. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Παδιώτη έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Uh, never mind. <laughs> Ε, ε, there are two points. Δύο πράγματα είναι σχετικά και πρέπει να γίνουν κατανοητά στη συγκεκριμένη αναφορά. Πρώτα απ' όλα είναι η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης. Αυτό είναι υποχρέωση που απορρέπει την οδηγία. Εν αυτή τη ενία, αυτή η απέτηση εφαρμογής σχεδίου δράσης που αναφέρεται στην αναφορά είναι κάτι που ισχύει. Όπως ήδη ανακοινώθηκε, η Οδηγία 2002-49 Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα μέτρα των σχεδίων δράσεως εφαρμόζονται σύμφωνα τη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων αρχών. Το ότι υπάρχουν οριακές τιμές είναι μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις που απαιτεί να, χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιηθεί η οδηγία όταν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Οι εθνικές αρχές αποφασίζουν όμως εάν και πότε και πώς θα παρέμβουν. Για τους σκοπούς της, περι... της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό θόρυβο, η οδήποτε μέτρο είναι αποδεκτό υπό την προϋπόθεση ότι συζητείται με τους πολίτες και υπό την προϋπόθεση ότι το σχέδιο υποβάλλεται εντός των συγκεκριμένων προθεσμίων προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επόμενο σχέδιο προβλέπεται για 18 Ιανουαρίου 2013. Προβλέπει δηλαδή η οδηγία εντός αυτής της προθεσμίας να ανα, επαναεξεταστούν, να ανασυνταχθούν τα σχέδια δράση που κανονικά ε, αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. Και κάτι άλλο που αναφέρεται στην αναφορά όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα των διαφόρων ισπανικών κανονισμών για τις οριακές τιμές. Ήρθαμε σε επαφή ανεπίσημα με τις ισπανικές αρχές σχετικά με αυτό, για να δούμε αν είναι βάσιμα αυτά που αναφέρονται και θα έρθουμε σε επαφή και επισήμω μαζί τους. 23 Φεβρουαρίου του 1996 ε, αυτή, ε, αυτός ο νόμος δεν εφαρμόζεται πλέον. Ισχύει ο γενικός νόμος, μας είπαν οι Ισπανικές αρχές. Συνεχίζονται οι συνομιλίες στις ανοιοκές αρχές. Θέλουμε να πούμε κατά πόσο μας ενημέρωσε σωστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Ισπανικές αρχές μας έστειλαν και άλλες πληροφορίες. Μας είπαν ότι το διάταγμα 3 του, 2003 ε, της ε, κυβέρνησης της Ανδαλουσίας καταργήθηκε από το διάταγμα 6 του 2012. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των ηχοπετασμάτων, προβλέπει οδηγία ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν για τα μέτρα τους. Αν αποφασίσουν τα κράτη-μέλη ότι αυτά είναι τα ενδεικνυόμενα μέτρα, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν παραβιάζουν τους κανονισμούς. Σας ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου. Πριν ξαναδώ στο άλλο στον κύριο Γκερέρο, υπάρχει συνάδελφο που ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Εγώ ως πρόεδρος ε, να πω, μάλλον πιο πολύ ως μέλος και όχι ως ε, προεδρεύων, ως μέλος της ομάδας μου, της ομάδας του ΕΛΚΑ να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δύο θέματα υπάρχουν το ένα το αναφέρει και εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παραβιάζονται διάφορε οδηγίε, άρα δικαίω ε, έχει καταθέσει την αναφορά του αναφέρον. Υπάρχει και κάτι άλλο που είπε ο αναφέρον, δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, ότι πριν από έξι μήνες ζήτησαν ε, απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχετε όμως απαντήσει μέχρι στιγμής. Έχετε λάβει γνώση των ισχυρισμών αυτών, των καταγγελιών αυτών που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί και αυτό ξέρετε είναι ανησυχητικό να μην έχουν λάβει δηλαδή απάντηση αυτές τις πληροφορίες που ζήτησαν οι αναφέροντες. Και επειδή στις 18 Ιανουαρίου 2013 θα τεθεί σε ισχύ μια νέα οδηγία, δεν ξέρω εάν πλέον μπορούμε να περιμένουμε την θέση ισχύ της οδηγίας αυτής. Δεν θα πρέπει να έχουν πάρει κάποια απάντηση αναφέροντες θα περιμένουμε τεθεί σε ισχύ η οδηγία. Θα ήθελα κάποιε απαντήσει από εσά. Ναι. Λάβαμε όλε τις πληροφορίε, τις έχω μαζί μου. Τις ξαναδιαβάσαμε. Δεν είδαμε νέες πληροφορίε όσον αφορά την οδηγία για περιβαλλοντικό θόρυβο, σύμφωνα με τις, ε, σε σχέση με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επειδή οι Ισπανικές αρχές υπέβαλαν πρόσφατα κάποιες πληροφορίες για την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων, ήθαμε σε επαφή μαζί τους ανεπίσημα και θα τους ρωτήσουμε. Εάν δεν έχουμε τελική απάντηση, όπως καταλαβαίνετε, από τις Ισπανικές αρχές, δεν έχει νόημα να πούμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε νέες πληροφορίες επίσημα για το θέμα. Όσον αφορά τις διάφορες οδηγίες, ζητώ συγγνώμη που ήμουν ασαφής. Δεν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες, αλλά μία οδηγία η Ευρωπαϊκή Οδηγία για, τον, για την Ιχορύπανση. Η προθεσμία 18 Ιανουαρίου 2013 είναι νέα προθεσμία για νέα σχέδια δράσης που θα πρέπει να εκπονηθούν από τα κράτη-μέλη. Και στην περίπτωση της αναφοράς ισχύει αυτό. Ήταν συμπληρωματικέ πληροφορίε αυτές που θέλαμε να δώσουμε στον αναφέροντα για να το εξηγήσουμε ότι υπάρχει και άλλη δυνατότητα με τη συμμετοχή των εθνικών αρχών να ζητηθούν άλλες δράσεις από τις εθνικές αρχές. Είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει και θα επαληθεύσει τα σχέδια δράσης και θα δει κατά πόσο τα σχέδια δράσης αυτά εγκρίθηκαν και θετήθηκαν εντός της ε, προβλεπόμενης ε, προθεσμίας. Επειδή είπατε ότι ερευνάτε το θέμα, συνεχίζετε να το ερευνάτε. Σας παρακαλώ λοιπόν να συνεχίσετε Οπότε πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά μέχρι να έχουμε την ενημέρωση από τις ε, έρευνες που όπως είπατε διεξάγεται. Ωραία. Θέλετε να πείτε τίποτα κύριε Γκερέρο, καταλήγοντας για το θέμα αυτό. Βεβαίως. Θα ήθελα να πω στον εκπρόσωπο της Κομισιόν ότι η οργάνωσή μας ξέρει ότι κάθε πέντε χρόνια πρέπει να γίνονται προγράμματα δράσης κατά των νέων θορύβων. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε για αυτό το διάταγμα 23 του 96 που το εφαρμόζουν κάποιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης ακόμη. Ευχαριστώ πολύ που συνεχίζετε να το μελετάτε, να το διερευνάτε. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Να περάσουμε στη 15 του κυρίου Ράνχαρντ Ούριχ, γερμανικής Ιθαγένειας, από πλευράς της ε, οργάνωσης ε, φίλη... Α, και αυτή πρέπει να αναβληθεί. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Τι θα γίνει. Υπάρχει καμιά άλλη που πρέπει να αναβάλουμε. Α, μόνο αυτή και η προηγούμενη. Α, ωραία. Οπότε θα συνεχίσουμε τώρα με τη 16. Ανα... όχι... Me dicen que ha vuelto el... Ωραία. Να περάσουμε στη 12. Αναφορά από πολίτη... Συγγνώμη, όχι, 13, 13. 306 Χάρμελ Σπιτέρι, Μαλτέζικης Ιθαγένες, ε, εξ ονόματος των κατοίκων της Σάντα Βένερα, 160 υπογραφές σχετικά με ισχυρισμούς για ρήπανση του αέρα και χορύπανση που περνούν τα όρια που θεσπίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ εξαιτίας περιφερειακής οδού στην περιοχή Σάντα Βενέρα όπου διαμένουν. Ο κύριος Γκασπαρινέτη θα μας ενημερώσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, με συγχωρείτε για θέση. Όσον αφορά αυτή την αναφορά. Ερεύνησε περαιτέρω η Επιτροπή και συμπεριλήφθηκε σε συμπληρωματική ε, ανακοίνωση αυτό. Κάθε χρόνο ξέρετε ότι ενημερούν τα κράτη-μέλη σχετικά με τα θέματα σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στις διάφορες περιοχές. Βάσει του οδηγία της Οδηγίας 2008 κάθετος 50 και όσον αφορά την ποιότητα του αέρα στη συγκεκριμένη στική περιοχή μπορούμε να συνοψίσουμε ότι είναι η εξή. Για τα αερούμενα σωματίδια PM10 σύμφωνα με την ορολογία της οδηγίας υπάρχουν ε, ναι, ετήσιες άξιες 30 ε, μικροσωμάτια ανακυβικό μέτρο και καθημερινή οριακή τιμή που δεν πρέπει να ξεπερνιέται πάνω 35 μέρες το χρόνο και σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών της Μάλτας η μερίσια τιμή ε, ξεπεράστηκε 37 ημέρες. Και μετά από τις φυσικές συνεισφορές που μπορούν να αφαιρεθούν σύμφωνα με την οδηγία, διότι η Μάλτα υπόκειται ε, σε συχνά φαινόμενα ανέμων που φυσούν από τη Σαχάρα και φέρνουν σκόνη από τη Σαχάρα. Μπορούν να αφαιρεθούν λοιπόν οι φυσικές συνεισφορές, όπως είναι ο άνεμος που φυσάει και φέρνει άμμο από την ε, έρημο, αλλά μετά αυτή την αφαίρεση και πάλι ξεπερανιούνται οι οριακές τιμές στην ε, Μάλτα. δεν είναι η πιο σοβαρή κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την ρήπανση ατμοσφαιρικού αέρα, διότι σε άλλες περιοχές της Ευρώπης οι υπερβάσεις είναι πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες, αλλά παραβιάζεται η οδηγία διότι πρέπει παντού να τηρούνται οι οριακές τιμές σύμφωνα με την οδηγία και εδώ έχουμε παραβίαση της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο. Ο κύριος Γιάννου. και πάλι ζητάει συγγνώμη ο κύριος Μπουσουτήλ που δεν μπορεί να είναι παρόν αλλά μου ε, έδωσε τις σημαντικές ερωτήσεις που ε, εξεπώνησε προς το συμφέρον και του αναφέροντος και της ουσίας. Ερώτημα του αναφέροντος. Θα ήθελα να μάθει εάν η ποιότητα του αέρα είναι εντός των ορίων της ε, κοινοτική και αν όχι, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ερώτημα λοιπόν προς την Κομισιόν, το κύριο. Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς το είπε ο εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής. Τηρούνται οι διατάξεις οδηγίας ή όχι. Γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν ξέρω να κατάλαβα καλά. Οι αρχές της Μάλτας λένε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές οξυδίων του αζότου. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που λένε το αντίθετο. Είναι σημαντικό, ε, όχι όταν χτίζουμε δρόμους να μην τηρούμε τις ε, διατάξεις. Να πω σαφώς ότι είναι κατανοητό ότι οι αναφέροντες λόγω της τόσο διαφορετικής πληροφόρησης έχουν ανησυχίες ε, για την υγεία τους. Έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Συγκεκριμένα ρωτάω την Επιτροπή πώς εκτιμά συνολικά την κατάσταση συγκεκριμένα. Τηρούνται οι οριακές τιμές ή όχι. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ισχύουν αυτά που ε, υπόθηκαν τελευταία ότι είναι εντός των ορίων ε, οι τιμές. Μπορεί να μας επιβεβαιώσει την πληροφόρηση. Ευχαριστώ κύριε Γιάννου, Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να εξηγήσω περαιτέρω τι είπα στην πρώτερη απάντηση. Αυτό που δεν είπα, διότι ήταν στη γραπτή μα ανακοίνωση, ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση που φαίνεται να είναι η πηγή των ανησυχιών για του αναφέροντε δυστυχώ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία IPPC 2008-1. Οπότε το περιθώριο ελιγμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσης και το τονίζω αυτό Ευρωπαϊκή Ενώσης διότι έχουμε και την ε, χώρια νομοθεσία, είναι περιορισμένη όσον αφορά τη συγκεκριμένη μονάδα. Όμω, η ποιότητα, οι οριακές τιμές του ατμοσφαιρικού αέρα που αναφέρονται στη 2008 2015 πρέπει να γίνονται σεβαστές ανεξάρτητα από τις πηγές ρήπανσης. Όποια και αν είναι η πηγή της ρήπανσης, είτε καλύπτεται η πηγή είτε δεν καλύπτεται από νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οριακές τιμές του ατμοσφαιρικού αέρα θα πρέπει να τηρούνται. Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει όσον αφορά τη συγκεκριμένη ζωνή όσον αφορά το PM10, όσον αφορά τα σωματίδια, τα ορούμενα σωματίδια, για να το μεταφράσουμε αυτό σε πιο εύληπτη γλώσσα. Οπότε προτιθέμε θα το θέσουμε στις αρχές της Μάλτα το θέμα, αυτό το μήνα πιθανότατα θα το αναφέρουμε και όσον αφορά το θέμα της συμμόρφωσης οριακής τιμές, ε, εν γέννη αυτό είναι οριζόντιο θέμα και η Μάλτα δεν είναι το μόνο κράτο μέλος που έχει υπερβάσει σε κάποιες περιοχές και αστικέ περιοχές και απαιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση κατ' όλων ή κατά κανενός, αλλά ιδεοδός θα έπρεπε ταυτόχρονα να κινηθούμε, να κινούμαστε ταυτόχρονα κατά όλων των κρατών μερών όταν υπάρχουν υπερβάσεις. Ευχαριστώ κύριος Γιάν και πάλι. Από ό,τι κατάλαβα, ο διάλογος μεταξύ Κομισιών και αρχών της Μάλτας δεν έχει ακόμη καταλήξει θα πρότεινα λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Βεβαίως, εάν δεν θέλει να πει κανείς ε, τίποτε άλλο, θα την κρατήσουμε ανοιχτή. 15 την έχει υποβάλει ο κύριος Κούρη από πλευρά τη οργάνωση φίλη της γης της Αυστρίας υπογραφές 98.500 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση τη πυρηνική ενέργεια που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι παρόν. Είναι παρόντες οι αναφέροντες. Α, ωραία. Θα δώσω το λόγο λοιπόν σε αυτούς. Μισό λεπτό. Ποιο θα μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την ε, Friends of the Earth της Αυστρίας όπως σας είπαμε, έχουμε πάνω από 8.500 υπογραφές. Θέλουμε να μιλήσουμε για την πυρηνική ενέργεια, διότι μετά τα ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της ε, Φουκουσίμα διαπιστώσαμε ότι η πυρηνική ενέργεια δημιουργεί ε, συνεχείς απειλές για την ε, ζωή των ανθρώπων και για μια ακόμη φορά είδαμε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής. Υπό το πρίσμα λοιπόν ε, των επιπτώσεων ε, της ε, καταστροφής της Φουκουσίμα ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την υποβολή αναφοράς. Θέλουμε να λάβει δράση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα ζητούμε σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών σταθμών. Πρώτα να κλείσουν οι πλέον επικίνδυνοι και σιγά σιγά να καταργηθεί όλη η στάθμη. Συγγνώμη που η φωνή μου είναι λίγο έχει κλείσει ο λαιμό. μου. Επίσης θέλουμε να αναπτυχθούν πηγές ανανεώσιμης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εφαρμοστούν μέτρα ενεργειακή απόδοσης ε, με καθαρά υλικά, αντικατάσταση των ορεικτών καυσίμων. Υπευλήθησαν λοιπόν πολλέ υπογραφές, 98.500 ε, από το Σεπτέμβριο 2011. 700.000 πολίτες είναι ενημερωμένοι πλέον για τις ε, επιπτώσεις της πυρηνικής ενέργειας και έχουν υπογράψει την αναφορά και ζητούν από του αιρετού εκπροσώπου να σεβαστούν τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Αυτό δεν, τα δικαιώματα αυτά δεν γίνονται σεβαστά όσο συνεχίζει να χρησιμοποιεί την πυρηνική ενέργεια, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει για θέματα ενέργεια να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη, όπω και την πυρηνική ενέργεια. Είμαι αυστριακή. Ε, η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών στη χώρα μου είναι αντίθετη προ την ε, πυρηνική ενέργεια. Πώ μπορούν να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματά μου όταν και στα σύνορα της χώρας μου ε, ένα πυρηνικό εργαστήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά υπάρχουν σε απόσταση 60 έως 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βιέννη πάνω από 10 ε, πυρηνικοί σταθμοί. Υποβλήθηκαν ε, στα τεστ αντοχής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαπιστώθηκε ότι απαιτούνται μέτρα τεχνικής αναβάθμισης των δραστήρων. Κανένας δεν τηρούσε τα πρότυπε, τι προδιαγραφέ ασφαλεία, λαμβάνοντα υπόψη ότι η δεν σταματάει στα σύνορα τα πολιτικά. Η απόφαση ενό κράτου μέλου να απέχει από την πυρηνική ενέργεια δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ε, πολιτών τη χώρα. Ε, με βάση τη συμβουλή που ακούσαμε, μπορεί να βασιστούμε στις αρχές τη προφύλαξης μεταξύ άλλων για να έχουμε την προστασία, να επιτύχουμε την προστασία της φύσης και για να μην ανεγερθούν οι πυρηνικοί ε, σταθμοί. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν ατυχήματα και έτσι θα δημιουργηθούν ε, κίνδυνοι για το περιβάλλον, τη βεπικιλότητα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη ζωή των πολιτών. Και αυτά είναι κατοχυρωμένα από τις συνθήκες δικαιώματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία, θα πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια για την κατάρριξη πυρηνική ενέργεια και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο και η Κομισιό να ακούσει τι φωνέ των πολιτών που ανησυχούν και να βρει έναν τρόπο να δημιουργήσει σχετική νομοθεσία ώστε να υπάρχει ένα καθαρό, ασφαλέ σύστημα για το μέλλον τη Ευρώπη. Ελπίζουμε στο μέλλον να μην ε, χρειαστεί μια ακόμη ε, καταστροφή για να καταλάβουμε όλοι μα ότι οι συνέπειε μια πυρηνική καταστροφή δεν μπορούν να θεωρούνται μόνο εθνικό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόλφαν Κίμπ από τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να τονίσω ότι η πυρηνική ασφάλεια, αυτονόητο είναι, έχει μέγιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε συμφωνούμε από αυτού του σημείου με τον ε, αναφέροντα. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι στα πλαίσια των συνθήκων. Η συνθήκη Ευρατών εξακολουθεί να ισχύει. Εκτός αν αναθεωρηθεί ή καταργηθεί. Το άρθρο 149, 194 συγγνώμη, καθορίζει ότι κάθε χώρα μπορεί να καθορίσει την ενεργειακή της πολιτική. Υπάρχουν πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου, υπάρχουν πρωτοβουλίες από πλευράς πολιτών που μπορούν να στραφούν προς την Κομισιόν για να αλλάξει αυτό το νομικό πλαίσιο. Αλλά όσο δεν έχει αλλάξει, εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να τηρείται. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη, όπως ε, ακριβώς το αναφέρει και ο αναφέρον, με βάση την σημερινή κατανομή αρμοδιοτήτων πρέπει να φροντίζουν για την ασφάλεια των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων. Συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας, εάν το επιθυμούν, να σταματήσουν τη λειτουργία μιας πυρηνικής εγκατάστασης. Την προηγούμενη εβδομάδα θα ακούσατε τον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την ενέργεια όταν παρουσίασε την ανακοίνωση για το κλείσιμο των ε, τεστ αντοχής Συνοψίζοντας, η ανακοίνωση τονίζει δύο σημεία. Ότι την πρωτοβουλία πρέπει να αναλάβουν και πάλι τα κράτη-μέλη για να εκπονήσουν τεχνικά σχέδια για την βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους και από την άλλη πλευρά βεβαίως πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε να εκπονήσει το γενικότερο πλαίσιο από πλευρά νομική ασφάλεια επίση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Ούτω ώστε να πιέσουμε να ενισχυθούν στι αρμοδιότητε και την αυτονομία του οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η Μάργαρετ. Η Μάργαρετ δεν ξέρω αν θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Όκεν αυτή η έκθεση του Έτιγερ ε, και εγώ ήθελα να την αναφέρω. Όλοι ανησυχούμε πολύ για την κατάσταση. Εμείς ως χώρα αποφασίσαμε στα μέσα της δεκαετίας του 80 να μην βασιστούμε, να μην έχουμε καθόλου πυρηνική ενέργεια μετά από μια συζήτηση που κράτησε δεκαετίες. Και ο λόγος δεν ήταν ε, το Τσερνόμπιλ. Η απόφασή μας λήφθηκε το 85, ένα χρόνο πριν βασίστηκε στο ότι δεν ήταν να τον εξασφαλίσουμε απόλυτα ασφαλείς πυρηνικές εγκαταστάσεις. Κοιτάξτε, οι ε, εταιρείε που ε, δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα μυρίζουν το χρήμα και ξέρουν ε, πώς να το ξετρυπώσουν. Αλλά, ακόμη και αυτές δεν ήταν σε θέση να μας πούνε ότι είναι αδύνατον να προκύψει πυρηνική καταστροφή και μας είπαν ότι αν υπάρξει πυρηνική καταστροφή δεν ήταν δυνατόν ποτέ να αποζημιώσουμε όσους μπορεί να φυγούν. Και αυτά μας τα είπαν και οι ε, εταιρείε ασφάλισης και αντασφάλισης. Και καταλαβαίνοντας λοιπόν ότι αν οι ασφαλιστικές εταιρείε που θέλουν να ασφαλίζουν, να βγάζουν φράγκα μας ε, ε διευκρίνησαν ότι δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν τότε και εμείς πιστήκαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια σχέδια. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Και τα σχέδια δράσης ούτως ή άλλως δεν είναι τους, η μόνη πρόσφατη ε, πυρηνική εγκατάσταση που έχει παραγγελθεί τα τελευταία 30 χρόνια είναι στην Φιλανδία και ακόμη δεν έχει τελειώσει, έχει καθυστερήσει, έχει υπερβεί το κόστος. Πρέπει λοιπόν ομού με τους πολίτες όχι απλώς να κρατήσουμε απλή την αναφορά, αλλά να τονίσουμε ότι για μας ε, δεν μετράει μόνο το χρήμα, αλλά η φύση και οι άνθρωποι. Ευχαριστώ Μαργαρίτ. Ο κύριος Ζίμπερτ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η πράσινη συναδελφός μου ε, ε, αναφέρθηκε τόσο πολύ στα χρηματικά θέματα. Συνήθω δεν περιμένουμε τέτοιου τύπου επιχειρηματολογία, αλλά νομίζω ότι είναι οι Δανέζικη μαζί με την πράσινη ψυχή σα που σα έκανε να εκφραστείτε έτσι. Υποστηρίζουμε αυτήν την ε, ε, αναφορά. Εγώ είμαι ε, νομομαθής. Όπως ξέρετε όπου υπάρχουν δύο νομομαθείς ε, υπάρχουν τρει απόψεις. Είναι πολύ σωστό λοιπόν να βασιστούμε στο 194 αλλά πρέπει να ερμηνευτεί σωστά αυτό το άρθρο διότι αν ε, αφήσουμε στο κράτος μέλος ε, κάθε απόφαση για την ε, ενεργειακή του πολιτική, τότε είναι δικό μας καθήκον να φροντίζουμε για την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων. Όπως ξέρετε, τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια είναι στα σύνορα των κρατών. Οπότε αν υπάρξουν ατυχήματα, θα υπάρξουν ε, τεράστιες διαμεθοριακές επιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτήν την πλευρά της ασφάλειας, γιατί όπως είπαμε είναι διαμεθοριακό θέμα και θα μπορούσαμε να, έχουμε, ε, να δημιουργήσουμε μια κοινοτική αρμοδιότητα για τέτοια θέματα διαμεθοριακής ασφάλειας. Βεβαίως, αυτά που έκανε ο κ. Σέτιγκερ είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση. Κατέδειξε σαφώς ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ούτε μία πυρηνική εγκατάσταση που είναι απόλυτα ασφαλής. Χρειάζονται όμως ε, περαιτέρω βήματα, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια κοινή υπηρεσία, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη που θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτήν την ε, μορφή ενέργειας, να δίνουν δυνατότητα σε άλλα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις ε, αποτιμήσεις της ασφαλείας των εγκαταστάσεων αυτών. Είναι σημαντικό λοιπόν να το καταλάβει αυτό η κοινή γνώμη και όχι τα κράτη-μέλη να κάθονται πάνω στο πυρηνικά του εργοστάσια και να μην επιτρέπουν να ε, συζητηθούν τα προβλήματα ασφάλειά του. Πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουμε την κατάσταση αυτή, ούτω ώστε εμπειρογνώμονε και από άλλα κράτη-μέλη να μπορούν να συμμετάσχουν. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε μεταξύ άλλων επειδή υπάρχει αυτό το διαμεθοριακό θέμα ασφάλειας πρέπει να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμα μια διαμεθοριακή αρμοδιότητα, ούτω ώστε μέχρι να σταματήσουν αυτά τα εργοστάσια να έχουμε δυνατότητα να ελέγξουμε την ασφάλεια που θα μπορούσε να έχει τόσο τρομερές επιπτώσεις. Φυσικά, για το κόστος, το κόστος της αποσυναρμολόγησης και το κόστος της αποθήκευσης των καυσίμων είναι πολύ σημαντικό θέμα και πολύ δυσχερές. Ξέρετε τι γίνεται στη Γερμανία. Προκύπτουν τρομερά έξοδα, τρομερές δαπάνες. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να προσπαθήσει να αποτιμήσει το κόστος του συνολικού κύκλου από την εξόριξη του ουρανίου μέχρι την ε, τελική ε, αποθήκευση ε, των αποβλήτων καυσίμων θα καταλήξουμε τότε σε εκτίμηση ότι είναι τεράστιο το κόστος αυτής της μορφής ενέργειας. Θα ήταν ε, σκόπιμο λοιπόν η Κομισιόν να είναι λίγο πιο θαραλέα να μας κάνει τέτοιες μελέτες για το συνολικό κόστος. Υπάρχουν κάποιες λύσεις μέσω των ασφαλιών. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία ασφαλιστική εταιρεία που θα ήταν ε, διατεθειμένη να αναλάβει ένα τέτοιο κίνδυνο γιατί το κόστος ε, των αποζημιώσεων θα ήταν τρομερό. Εάν παραμείνουμε σε αυτές τις ε, κλασικές ε, ε, μεθόδους σχάσης, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι περιορισμένο το κάψιμο που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να περάσουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μην εμένουμε σε μια εντό εισαγωγικών πεπαλαιωμένη και επικίνδυνη μορφή ενέργειας. Καλωσορίζω λοιπόν την Επιτροπή και ελπίζω η Κομισιόν να συνεχίσει να ασχολείται με αυτήν και να απαντήσει στις ανησυχίες του αναφέροντος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζέμπερ. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρει κάτι από αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, Ευρωβουλευτές για τις παρατηρήσεις. Συμπληρωματικά, τα εξής. τα τεστ αντοχής που μόλις κάναμε, οι ομάδες μας, που ήταν ομάδες όπου διάφοροι εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες ε, εκτιμούσαν ένα στα αποτελέσματα του άλλου, με τη συμμετοχή της Κομισιόν. Δεύτερον, για την ε, αντιμετώπιση των αποβλήτων υπάρχει οδηγία από πέρυσι για την αντιμετώπιση των ενεργών αποβλήτων. Όλες ε, οι χώρες μέλη και όλοι Όλε οι εταιρείε που ασχολούνται με αυτά, όλε οι πυρηνικέ καταστάσει πρέπει να ασχολούνται και με την αντιμετώπιση των αποβλήτων του. Και ε, τρίτον, δεν μα ενδιαφέρει μόνο η τεχνική ασφάλεια, αλλά μα ενδιαφέρει και το θέμα τη ε, αστική ευθύνη. Συμπεριλαμβανομένων και των τροφίμων που μπορεί να απολυθούν ραδιενεργώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε... Σα ευχαριστώ. Ο αναφέρον ή αναφέρουσα στην προηγούμενη περίπτωση, σα δίνω δύο λεπτά αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Θέλω να πω ότι θα εξακολουθούμε να θέτουμε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω όλων των δημοκρατικών διαθεσίμων μέσων και θα υποβάλουμε και Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σχετικό αίτημα. Μάλιστα. Η Μάργαρετ ε, μόλις που το άκουσε και Έσκασε χαμόγελο. Τη αρέσει πάρα πολύ όταν ακούει για πρωτοβουλίε πολιτών. Ωραία, αν συμφωνείτε λοιπόν, όπω είπε και ο κύριο Ζέμπερ, διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά. Κύριε Ζέμπερ, κύριε Άουκεν. Βεβαίω, να παραμείνει ανοιχτή. Πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει λοιπόν. ευχαριστήσω τους αναφέροντες για την παρουσία τους εδώ και τώρα πηγαίνουμε στην αναφορά 1078 του Ιωσέμπα Μίρεν Σάινς Δελαγέρα Εγκαρτσία Ισπανικής Ιθαγένειας σχετικά με το σταθμό πυρηνικής ενέργειας της Γαρόνια στο Μπούργος. Δεν ξέρω αν έχει έρθει πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, είστε πάλι εσείς ε, αρμόδιος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο πυρηνικός σταθμός αυτός στο Μπούργκος μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι τον Ιούλιο του 2013. Δεν ζητήθηκε παράταση της άδειας λειτουργίας του, οπότε το επόμενο καλοκαίρι θα λυθεί το θέμα. Ε, ναι, πράγματι. Υπάρχει κάποιο σχόλιο. Ο Βίλι Μέγερ. Το περίμενα ο κύριος Μέγερ. Ήθελα απλά να σχολιάσω ότι μέχρι να κλείσει ο πυρηνικός αυτοσταθμός πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και αναφορά. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της πυρηνικής ενέργειας. Ελπίζουμε λοιπόν πράγματι να μην υπάρξει παράταση στη λειτουργία αυτού του σταθμού. Και πρέπει να επαγρυπνούμε να μην ζητήσει παράταση η εταιρεία αυτή. Και πραγματικά ε, καλό είναι να επαγρυπνούμε και να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Πρόεδρος, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει παράταση, όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και όπως είπες και εσύ θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, να παρακολουθούμε τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία που λύγει ουσιαστικά ε, η άδεια λειτουργίας. Θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και εμείς. Περνάμε τώρα λοιπόν ε, στο σημείο 17 της ημερήσια διάταξη αναφορά 1026 του Γκρέντο Φέρστερ, Γερμανική σταγέννη σχετικά με την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στη θάλασσα. Είστε ο ειδήμων για αυτά τα θέματα, από ό,τι κατάλαβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, ναι, πράγματι. Όσον αφορά την αναφορά αυτή, εδρεύεται επί άρθρου που εμφανίστηκε στο Spiegel Online. Αν όντω έτσι είχαν τα πράγματα, αν ένας πυρηνικός σταθμός κατασκευαζόταν στη θάλασσα, τότε, σύμφωνα με το άρθρο 41 της συνθήκης Euratom, αυτό θα έπρεπε να καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό δεν ισχύει. Αν υπήρχε ένας υποθαλάσσιος πυρηνικός σταθμός, θα έπρεπε να καταχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 Ευρατόμ. Και ούτε αυτό έχει γίνει. Οπότε δεν μπορώ να προβώ σε σχετικές δηλώσεις, παρά να αναφερθώ στο θεωρητικό νομικό πλαίσιο για όλα αυτά. Να Θέλει κάποιος το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Όχι. Ουδής. Άρα, όπως μας πήγε ο εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα κλείσουμε την αναφορά αυτή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στην αναφορά περιθμών 18 που αφορά την επέκταση του πυρηνικού σταθμού του Τέμιλη στην Τσεχική Δημοκρατία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και πάλι. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ο συνάδελφός μου από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Να έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο αλλά επειδή μας τα λέγατε τόσο ωραία, θα συνηθίσαμε. Ο εκπρόσωπος ε, που πρέπει να μας μιλήσει αυτό το θέμα παρίσταται, ναι. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω στα αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διαδικασία της ανάλυσης όλων των ε, πληροφοριών που έστειλαν οι καταγγέλλοντες πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει και διαδικασία διαβούλευσης σε εξέλιξη για το εν αυτό έργο. Η Επιτροπή λοιπόν αναλύει τις πληροφορίες προς το παρόν και βέβαια προσέχουμε, επαγρυπνούμε για τα όσα συμβαίνουν σε ό,τι αφορά με την ανάπτυξη όλα τα υποχρεωτικά στάδια το οποίο πρέπει να επιτελέσουν οι αρχές για την ε, τήρηση της οδηγίας ε, για την ε, εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θέλουμε να σχετίσουμε αυτό το ζήτημα με τη διαδικασία ΕΠΕ και να μιλήσουμε και για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Στο άρθρο 4, παράγραφος 7, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη ουσιαστικά να μην παραβιάζουν την οδηγία, αλλά θα πρέπει να προϋποθέσουν να, να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις που συνοψίζονται στα εξής. ότι πρέπει να λαμβάνουν τα πρακτικά μέτρα για να πεντριάσουν τον, α, τις αρνητικές επιπτώσεις ε, στην ποιότητα των α, θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση εκ του σύνεγγης, θα προσέχουμε για να διαπιστώσουμε κατά πόσον τηρείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου αυτού. Ευχαριστώ. Έχει κανείς σχόλια. Α, ο κύριος Ζήμπερτ. Θέλω να μιλήσω για τα θέματα που αφορούν τα ύδατα στο άρθρο 4. Ε, προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες ε, παρεκκλήσεις αλλά τονίζει ότι μόνο σε συγκεκριμένε περιπτώσει μπορούν να υπάρξει μια χαλάρωση. Αρμόδιε είναι οι εθνικέ αρχέ. Η Κομισιόν πρέπει να ελέγξει εάν έχει τηρηθεί αυτό ο κανόνα, να εξετάσει συγκεκριμένα εάν και κατά πόσο λόγω της θέρμανσης αυτών των απορρίψεων υδάτων μπορεί να υπάρξουν μεγάλες ε, ε, βλάβες στο περιβάλλον. Και δεν νομίζουμε ότι έχει να κάνει με αυτό το ε, σοβαρά τροποποιημένο σώμα ύδατος. Πρέπει λοιπόν να παρατηρήσει την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και άλλα θέματα ασφάλειας, αλλά δεν αναφέρονται σε αυτή την αναφορά, αλλά πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν συνεχώς ε, βλάβες σε αυτό το πυρηνικό σταθμό που δεν αναφέρονται ή αναφέρονται με καθυστέρηση. Γι' αυτό θα έπρεπε η Κομισιόν να παρακολουθεί αυτόν τον πυρηνικό σταθμό ούτως ώστε να ε, επιβάλλει την τήρηση όλων των ε, διατάξεων ασφάλειας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ζίμπερτ Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Η κυρία Ντέμελιν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Μόλις πρόλαβα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα να είμαι παρούσα. Συμφωνώ με τα επιχειρήματα του κυρίου Ζίμπερτ και με το αίτημά του προς την Κομισιόν. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θα πρέπει να εξεταστεί συγκεκριμένα, να λάβετε σοβαρά αυτή την απαγόρευση επιδείνωσης της κατάστασης γιατί το Τέμελιν είναι παράδειγμα εγκατάστασης όπου δεν έχουν γίνει επαρκώς μελέτες, δεν έχουμε παρακολουθήσει επαρκώς την κατάσταση. Είναι λοιπόν σαφής η κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε αναχείρα στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, να δούμε πώς εφαρμόζουν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις ε, τις διατάξεις της δεν πρέπει να υπάρξει επίοικια, είναι θέμα ποιότητας των υδάτων. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία εκπρόσωπος της Κομισιόν θέλει να μας πει τίποτα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζίμπερτ για τα σχόλιά του. Τα εκτιμώ ιδιαίτερα. Πρόκειται λοιπόν για την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και μία εξαίρεση από το 4-7. Τα κράτη-μέλη όταν ετούνται εξαιρέσεων. Πρέπει να παρακολουθήσουν, να εφαρμόσουν πολύ προσεκτικά όλα τα βήματα της οδηγίας για το πώς χορηγείται αυτή η εξαίρεση. Παρακολουθούμε τα διαχειριστικά σχέδια που μας έχει υποβάλει η Τσεχική Δημοκρατία από αυτού, ούτως ώστε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η χώρα αυτή να υποβάλει με τον ορθό τρόπο, εάν θεωρούν ότι ε, ε, ε, υπάρχει περιθώριο εξαίρεση με βάση το άρθρο 4,7. Θαυμάσια λέει ο πρόεδρο. Θα ε, τη, ε, κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, αναφορά μέχρι να λάβουμε πληροφορίε από τι τσεκέ αρχέ. Με ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει πρόσωπο τη Κομισιόν για τι δύο επόμενε αναφορέ, 19 και 20. Οπότε δυστυχώ θα πρέπει να αναβληθούν. Η 21 όπως ξέρετε, θα συζητηθεί με παρουσία του Αντιπροέδρου Τατζάνη, που προβλέπεται για τις 11.30 περίπου. Οπότε θα αναβάλουμε μέχρι τις 11 παρατέταρτο. Μέχρι τις 11 παρατέταρτο. Για να είναι παρόν παρόντα όλα τα άτομα που θα πρέπει να είναι παρόντα. Ευχαριστούμε. Μέχρι τις 11 παρατέταρτο, ελπίζοντας να είναι εκπρόσωποι της Επιτροπής, διότι αναφέρονται στην εδώ μέχρι τις 11 παρατέταρτο. 11 παρατέταρτο. Αντώνη. Να, Please, Σας παρακαλώ συνάδελφοι να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε συγγνώμη λοιπόν για αυτή τη διακοπή. Μπορούμε να ξεκινήσουμε εκ νέου για με 429 του κυρίου Ρόμπερτ Χουλστόν που είναι παρόν. Μέχρι το λόγο. Ευχαριστώ κ. Ευχαριστώ που το θέσατε στην υπηρεσία σας διάταξη. Κυρία Πρόεδρε, είναι λίγο απογοητευτικό ότι η αναφορά μας που υποστηρίζεται από 7.000 υπογραφές υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο πριν από 2,5 χρόνια και δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος έκτοτε επί του θέματος. Ελπίζω η σημερινή μας συνεδρίαση να δώσει μια όθηση στην ε, περάτωση της διαδικασίας ε, λήψης της αναγκαίας ενημέρωσης από τις ε, Ισπανικές Αρχές, ούτως ώστε η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να λάβουν θέση για την νομοτυπότητα της διαδικασίας να κατασκευαστούν 1.500 νέες κατοικίες στο τελευταίο τμήμα της Οριουέλα Κώστα. Η αρχές της Οριουέλα περιμένουν το Κοινοβούλιο μέχρι τις 5 ε, Νοεμβρίου. Να σας διαβάσω δύο παραγράφους από ένα ψήφισμα που ενεκρίθη από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Οριουέλα τον περασμένο Μάιο για να καταστεί σαφές ότι η Οριουέλα παραμένει, περιμένει τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών. Η πρώτη, παράγραφος που μας ενδιαφέρει, θα τη διαβάσω ισπανικά, επαναλαμβάνει προς το Υπουργείο Εξωτερικών την ε, πρόθεσή μας, την, ε, το ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναθεωρήσουμε και να εφαρμόσουμε τα μέτρα που θα θεωρηθούν αναγκαία από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβανομένης της αναβολής της, ε, της εκτέλεσης του έργου παρακαλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβαλλοντικών Θεμάτων να καθορίσει επιγόντως τις ενδεχόμενες παραλήψεις στη μεταγραφή των ευρωπαϊκών οδηγιών ούτως ώστε ο Δήμος της Οριουέλα να μπορέσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα στα πλαίσια του νόμου. Αυτές οι ε, σημαντικές παράγραφοι εγκρίθηκαν από όλα τα κόμματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Οριουέλα όταν συνεδρίασε το Μάιο εν Ολομελία. Είναι πολύ σημαντικό κυρία Πρόεδρε να λάβει θέση η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για το εάν και κατά πόσο είναι νομότυπο αυτό το πρόγραμμα οικοδόμησης κατοικιών με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επειδή ε, πιστεύω ότι δεν είναι νομότυπο, δεν ε, ε, συμμορφούνται προς την ε, ενωσιακή νομοθεσία. Θα υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα να επανυποβληθεί αυτό το σχέδιο, ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι πολύ πιο αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες που έχουν τεθεί σε ισχύ τα τελευταία 25 χρόνια από τότε που υπήρξε η πρώτη έγκριση για αυτό το κατασκευαστικό σχέδιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τις αρχικές σας σκέψεις, να πω ότι από όταν υπευλήθη η αναφορά, η Επιτροπή Αναφοράν υπέβαλε έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει πληροφορίες. Έδωσε μια πρώτη απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μερική όσον αφορά αρμοδιότητες και έστειλε και έτοιμα στις Ισπανικές Αρχές για κάποια ενημέρωση. Αυτό το, αυτό το 1,5 έτος δεν πέρασε εις θα ακούσουμε νέες πληροφορίες τώρα εκ μέρους του υπευθύνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα πάρει το λόγο, ο κύριος Ράμος Φλόριντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, όταν υποβλήθηκε αυτή η αναφορά και ε, τη λάβαμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες ε, της Επιτροπής την ε, μελέτησαν με βάση το νοσιακό δίκαιο για το περιβάλλον που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για αυτή την περίπτωση για να δούμε αν υπήρχε ενωσιακή αρμοδιότητα. Οι οδηγίες, όπως ε, εξηγήσαμε στην ενημέρωσή μας προς το Κοινοβούλιο που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, για αυτό το σχέδιο είναι από τη μία οι οδηγίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι ΆΒΕΣ και οι Habitat, και Θέλαμε να δούμε συγκεκριμένα εάν θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το Natura 2000, το δίκτυο. Επίσης έχουμε την οδηγία του 85, που αυτή τη στιγμή είναι η οδηγία 2011 κάθετος 92, η οποία οδηγία απαιτεί να υπάρξει ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για συγκεκριμένα έργα. Όπως ξέρετε, τα πρόγραμμα του παραρτήματος 1 πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν σε μελέτη επιπτώσεων, ενώ όσες είναι στο παράρτημα 2, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, με τις διαστάσεις του έργου και με τα κριτήρια που έχει καθορίσει το κράτος μέλος κατά τη μεταγραφή της οδηγίας του εθνικού δίκαιου, μπορούν λοιπόν να μελετήσουν κατά περίπτωση οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβουν περισσότερη πληροφόρηση εκτό από αυτά που μα έστειλε ο αναφέρον, τον οποίο ευχαριστούμε. Απευθύνθηκαν στι ισπανικέ αρχέ που ήταν αρμόδιες για το θέμα αυτό. Υπήρξαν τρει ε, ανταλλαγέ ε, πληροφοριών μεταξύ Κομισιών και Ισπανικών Αρχών. Στην πρώτη αρχική μα αίτηση, επειδή δεν είχαμε επαρκή πληροφόρηση, στην απάντηση ζητήσαμε δεύτερη φορά και φέτο τρίτη φορά ενημέρωση. Πώς έχει τώρα η κατάσταση. Οι Ισπανικές αρχές σε πρώτη φάση υποστήριξαν ότι αυτό το σχέδιο κατασκευής 1.500 κατοικιών στην παράκτια περιοχή του Οριουέλα της επαρχίας του Αλικάντε ενεκρίθη από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο του 2007. Οι Ισπανικές αρχές αναγνώρισαν ότι δεν είχε υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποστήριξαν ότι αυτή η περιοχή ήταν περιοχή όπου μπορούσε να υπάρξει δόμηση με βάση το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο για την περιοχή το οποίο εκπονήθηκε το 1984. Οι Ισπανικές Αρχές λοιπόν στην αρχή είπαν ότι η οδηγία για την ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, γιατί υπήρχε ένα γενικό σχέδιο χροταξία που είχε εγκριθεί πριν από την ε, θέση σε ισχύ τη οδηγία. Και μα είπαν επίση ότι το δίκτυο Natura 2000 δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από αυτέ τι κατασκευέ, διότι στην περιοχή, η περιοχή αυτή δεν περιλαμβάνεται στο δίκτυο. Είναι κοντά μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 που δεν θα επηρεαζόταν λοιπόν από αυτές τις κατασκευαστικές εργασίες. Επίσης, οι ισπανικέ Αρχές είπαν ότι παρά όλα τα προηγούμενα, η Γενική Διεύθυνση της Κοινότητας της Βαλένθια, που είναι αρμόδια, έλαβε μια σειρά μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις αυτού του έργου στο περιβάλλον. Πώς έχει τώρα η κατάσταση. Μας ενημέρωσαν οι ισπανικέ αρχέ, ότι έχει αναβληθεί η εφαρμογή του, έχει μπλοκαριστεί και σε μία από τις ε, μεταγενέστερες απαντήσεις τους μετά την ανταλλαγή αυτή και το αίτημα πληροφόρηση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να σας ε, ενημερώσουμε ότι οι Ισπανικές Αρχές δεσμεύτηκαν να κάνουν ένα screening, δηλαδή μία μελέτη του προγράμματος αυτού, για να δουν εάν και κατά πόσο θα έπρεπε να υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή είναι η νομική υποχρέωση που, όπως είπα στην αρχή, απαιτεί η οδηγία για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή τροποποίησαν οι Ισπανικές αρχές την αρχική του θέση όπου έλεγαν ότι δεν εφαρμόζεται εδώ αυτή η οδηγία και ναι δεν αναγνωρίζουν τώρα το αντίθετο αλλά είναι διατεθειμένες να κάνουν ένα screening, να κάνουν μια μελέτη όπως ακριβώς την απαιτεί αυτή η οδηγία. Η τελευταία απάντηση των Ισπανικών αρχών μας ενημέρωσε ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία screening και οι περιφερειακές περιβαλλοντικές αρχές απευθύνθηκαν σε διάφορες ε, οργανώσεις ε, για να λάβουν την άποψή τους, για να κάνουν τις αναγκαίες διαβουλεύσεις που ε, είναι τμήμα κάθε διαδικασίας τέτοιου screening. Επίσης, οι δημοτικές αρχές της Όριουέλα δεσμεύτηκαν να μην δώσουν τις αναγκαίες δημοτικές άδειες για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο που όπως σας είπα αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένο μέχρι ότου ολοκληρωθούν αυτές οι περιβαλλοντικές διαδικασίες. Όπως είπε και ο κύριος Αναφέρον, το Δημαρχείο δήλωσε ότι είναι διατεθειμένο να κάνει όλες τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αποτιμήσεις. Οπότε, καταλήγοντας, μπορώ να σας πω ότι με βάση την ενημέρωση που έχουμε λάβει, οι διάφορες ισπανικές αρχές που είναι αρμόδιες σε επίπεδο αυτόνομη περιεφέρειας αλλά και σε επίπεδο Δήμου έχουν τροποποιήσει την αρχική του θέση. Λαμβάνουν λοιπόν τα μέτρα ούτω ώστε να εφαρμοστεί το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο που θα μπορούσε να ισχύσει σε αυτήν την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εσά. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Κοιτάξτε, θα μιλήσω δανέζικα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό, να το παρακολουθεί κανείς. Οι Ισπανικές αρχές ξαφνικά θεωρούν ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση. Και υπάρχουν δύο πράγματα που με ανησυχούν και με ανησυχούν αρκετά. Σταμάτησε η κατασκευή, καλό αυτό. Αυτό όμως λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν σταματήσει πολλές οικοδομές. Και διαρωτώ με, οι ανησυχίες για το περιβάλλον σταμάτησαν την οικοδομή ή η οικονομική κρίση. Είχε γίνει σε άλλη περίσταση μια επίσκεψη στην... Εξετάσαμε τον αυτοκινητόδρομο Y30 και οι Ισπανικές αρχές τότε είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών. Για, το ονόμασαν, ε, αυτό το δρόμο οδό, ενώ ήταν φανερό ότι ήταν αυτοκινητόδρομος. Γιατί μια απλή οδός δρόμου, ε, οδός συγγνώμη πόλης, δεν υπόκειται στις απαιτήσει για ε, περιβαλλοντικές, περιβαλλοντικών συνεπειών. Αυτοκινητόδρομος όμως ε, εμπίπτει σε αυτήν την περίπτωση. Με ανησυχεί το ότι αποφασίζουν οι Ισπανικές αρχές ε, κατά πόσο ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία ή όχι. Έχω κακή εμπειρία από την Ισπανία. Εγώ κατάλαβα ότι ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να γίνει ε, αξιολόγηση περιβαλλοντικών συνεπειών και δεν εναπόκειται στις Ισπανικές αρχές κατά πόσο πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση ή δεν πρέπει θα πρέπει να γίνει και να συμμετάσχουν και οι πολίτες της περιοχής. Πρέπει να εισακουστεί η άποψή τους. Λοιπόν, εγώ προτείνω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να εκφράσουμε και την ικανοποίησή μας διότι άλλαξε η προσέγγιση, η κοινοτροπία και ελπίζω να υπάρχουν πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν, γνήσιοι λόγοι που οδήγησαν αυτή την αλλαγή και όχι άλλα στοιχεία. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω θετικά. Το θετικό είναι ότι οι επανειλημμένες ε, ερωτήσεις ε, της Κομισιόν έκαναν τις Ισπανικές Αρχές να αναγνωρίσουν ότι πρέπει να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών εκτόσεων και γίνεται και ότι επίσης σταμάτησε το σχέδιο αυτό. Το ερώτημα που πρέπει να συζητήσουμε βεβαίως είναι πώς λειτουργεί η ενημέρωση και η επικοινωνία γιατί από ό,τι κατάλαβα το Δημοτικό Συμβούλιο το ενέκρινε το 2007 και οι παραπάνω αρχές δεν ασχολήθηκαν με το αν θα έπρεπε να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπλώσεων. Έχω υπάρξει και εγώ τοπικά εκλεγμένος και όταν ε, εξετάζω ένα σχέδιο και αν δεν μου λέει κανείς παραπάνω ότι πρέπει να κάνω περισσότερα, τότε δεν κάνω τίποτα περισσότερο. Καταλαβαίνω λοιπόν τι έκαναν οι δημοτικές αρχές, κατανοητό, εφόσον ε, οι ισπανικές αρχές δεν συνεργάζονται καλύτερα, γιατί έχουμε μια ομάδα εργασίας ε, ως Επιτροπή Αναφορών για τις ισπανικές ακτές και εκεί διαπιστώσαμε ότι έχουν οικοδομηθεί ε, κάποια κτίρια σε λάθος μέρος. Δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος για την προστασία των ισπανικών ακτών προς το συμφέρον των πολιτών και το αναφέροντος βεβαίως είναι σημαντικό και διαμαρτύρομαι διότι εγώ πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο όντως φύγει το δίκτυο Natura. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άλλοι μπορεί να αγοράσουν ένα σπίτι και μετά από 10 χρόνια να διαπιστώσουν ότι το σπίτι τους βρίσκεται σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να έχει χτιστεί τίποτα. Κάτι λοιπόν μέχρι στιγμής ε, κατάφερε η αναφορά. Μας είπατε ότι σταμάτησε η οικοδόμηση. Γιατί σταμάτησε. Είναι μόνιμη αυτή η απόφαση να ανασταλεί ε, η οικοδομή αυτή ή είναι κάτι προσωρινό. Ποια είναι τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ. Ο αναφέρον για μια να δευτερολογήσει. Thank This has been very interesting. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων και άκουσα και τις απόψεις των βουλευτών της Επιτροπής σας. Θα τις μελετήσω με πολύ μεγάλη προσοχή και θα τα μεταφέρω στην Οριχουέλα και σημειώνω το ενδιαφέρον σας, τις προσπάθειες ε, που έχουν γίνει. Να σας πω, έχουμε συλλέξει ήδη 7.000 υπογραφές και αυτό δείχνει ότι οι πολίτες πραγματικά ανησυχούν, ανησυχούν για αυτό το project, για αυτό το έργο. Και ανησυχούν για το ότι θα επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον. Άκουσα με ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει μια αλλαγή στάσης από την πλευρά των Ισπανικών αρχών. Κατά την άποψή μου αυτό είναι ελπιδοφόρο και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μια τελική αξιολόγηση της κατάστασης. Δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα καλά. Οι αλλαγές, αυτή η αλλαγή στάσης, τι συνεπάγεται ότι οι Ισπανικές αρχές έχουν αποδεχθεί ότι θα υπάρξει εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή απλώς σημαίνει ότι τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τέτοια ΕΠΕ, ενώ κατά το παρελθόν έλεγαν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Το είπαν και οι αξιότιμοι βουλευτές. Δεν είναι σαφές πώς έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας το διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ για να απαντήσω στις ερωτήσεις τόσο των βουλευτών όσο και του αναφέροντος, να πω πρώτα απ' όλα ότι στο ερώτημα για ποιους λόγους έχει παραλύσει, έχει μπλοκαριστεί το έργο, αν αυτό είναι λόγω της δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οικονομικού, ε, Ευρωπαϊκού, ή λόγω της η απάντηση είναι ότι οι Ισπανικές αρχές δεν μας ε, κοινοποίησαν το λόγο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι και οι δύο και τα δύο αίτια. Σίγουρα όμως ε, και η αναφορά κινητοποίησε τις ισπανικές αρχές και επανεξέτασαν το ζήτημα αυτό, όπως και άλλα έργα πολεοδομικά, έτσι και αυτό αντιμετωπίζει τώρα πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Ό,τι αφορά τώρα την ε, κατάσταση, την τρέχουσα κατάσταση, οι Ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία του screening. Ποια είναι όμως ε, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν μετά αυτό το screening δεν τα γνωρίζουμε, δεν μας τα κοινοποίησαν για να δούμε κατά πόσον ε, θα γίνει πλήρης αξιολόγηση επιπτώσεων περιβαλλοντικών ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία που έχει εγκριθεί από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα προβλέπει ότι για τα έργα παραρτήματος 2, όπως είναι ένα τέτοιο πολυοδομικό έργο, απαιτείται η εκπόνηση αυτού του screening για την εφαρμογή των κριτηρίων τα οποία προβλέπονται από την οδηγία μετάταξη στο εθνικό δίκαιο. Αυτό, σε αυτή τη φάση βρίσκονται οι Ισπανικές αρχές αυτή τη στιγμή. λαμβάνουμε υπόψη και τα χαρακτηριστικά και τη θέση του project και τα κριτήρια που αναφέρονται για να δούμε κατά πόσον ε, θα πρέπει να υποκληθεί σε πλήρη διαδικασία, διαδικασία το έργο αυτό. Βέβαια, η πλήρη διαδικασία ε, αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ό,τι καλύτερο και για το περιβάλλον αλλά και για τη συμμετοχή των πολιτών, να μπορούν δηλαδή μέσω των διάβλων δημόσια ενημέρωση να εκφράζουν τι ανησυχίε του και τι παρατηρήσει του σε σχέση με αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή η αναφορά παραμένει ανοιχτή εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων. Ευχαριστώ εκ νέου τον αναφέροντα που μας επέστησε την προσοχή επί του θέματος. Πηγαίνουμε στην αναφορά του σημείου 20. Η αναφορά επιβλήθη από τον κύριο Πάτρικ Κούλεν που κατέγγειλε το 2006 ενδεχόμενη ρήπανση που προξενείται από μια χαλιβουργία και θεωρούσε ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος από την Ιρλανδική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος. Αυτή η αναφορά εξετάστηκε, ε, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες, υπήρξαν οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από την έρευνα η Επιτροπή των Αναφορών αποφάσισε να αρχιοθετήσει την αναφορά για έλλειψη, λόγω έλλειψης στοιχείων που υποστήριζαν τη θέση του αναφέροντος. Όταν ζητήθηκε και αρχιοθέτησε, ο αναφέρον παρουσίασε νέα στοιχεία όμως, το 2011, ζητώντας ε, να γίνει περαιτέρω επαλήθευση, να συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία και διερευνώντας η Επιτροπή μας το θέμα, και έστειλε και το κατάλληλο επίσημο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτή τη νέα φάση στην οποία μπήκαμε, στις 17 Φεβρουαρίου του 2012 λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πρώτη απάντηση που μας έδωσε εννέα στοιχεία και μας έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία όσον αφορά την καταγγελία για το ενδεχόμενο ρήπανση και για τις ευθύνε τη εταιρεία. Θα ακούσουμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι ο αναφέρον δεν είναι παρόν, ούτω ώστε να μα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένω νέα στοιχεία όσον αφορά την όλη διαδικασία που γίνεται για την εξακρίβωση αυτών των στοιχείων. Η κυρία Γκαμπριέλα Γκερζέντη είναι η πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητώ συγγνώμη γιατί σίγουρα δεν έχω προφέρει σωστά το όνομά της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας δώσω εν συντομία τα πιο σύγχρονα στοιχεία όσον αφορά το θέμα. Με βάση το ιστορικό παρουσιάσατε, οι πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας έχουν δοθεί στο Κοινοβούλιο. Ήρθαμε σε επαφή μετά εκ νέου με τις Ιρλανδικές Αρχές και ζητήσαμε διευκρινήσεις επί του θέματος. Επιβεβαιώθηκε βασικά ότι καλύπτεται η κατάσταση από την οδηγία περί και από την οδηγία IPPC. Αλλά δεν έχουμε λάβει ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την φύση των αποβλήτων που υπάρχουν, αν είναι επικίνδυνα τα αποβλήτα παράγονται ή δεν είναι επικίνδυνα. Και χρειαζόμαστε και άλλες διευκρινήσεις όσον αφορά την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της ε, ερυθράς λάσπης. Έχουμε ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στις Εθνικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EU Pilot, και πήγαμε στην Ιρλανδία Μάλλον δώσαμε στην Ιρλανδία αρχές Σεπτεμβρίου τις πρόσφατες πληροφορίες και ζητήσαμε διευκρινήσεις. Ποια είναι η φύση των αποβλήτων, θέλαμε να ξέρουμε, διότι αναλύσαμε το μεταξύ τις πληροφορίες που μας δόθηκαν από την ετήσια έκθεση, από τις ετήσιες εκθέσεις της εταιρεία. Δεν είχαμε πιο πριν αυτές τις πληροφορίες και από αυτές τις πληροφορίες μπορέσαμε να δούμε ότι είναι επικίνδυνα τα απόβλητα που παράγονται με βάση κάποια κριτήρια όσον αφορά την οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα και λαμβάνοντας υπόψη το ότι αν τα απόβλητα είναι υγρά ή αν είναι λάσπη που εμπεριέχουν μέταλλα ή συστατικά μετάλλων, αυτά τότε θεωρούνται απόβλητα επικίνδυνα. Και η ίδια οδηγία αναφέρει και το διαβροτικό χαρακτήρα που ε, μπορεί να έχουν τα απόβλητα που τα κάνει επικίνδυνα. Ε, και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο θέσαμε εκ νέου στην Ιρλανδία, θέσαμε το ερώτημα και θέλουμε και επιβεβαίωση και αποσαφήνιση για τη μέθοδο ξηράς αποθήκευση όπως αποκαλείται. Δηλαδή το περιεχόμενο ε, ε, του ε, υδροξιδίου του, του νατρίου αφαιρείται. Αν μας επιβεβαιώσει ότι είναι πραγματικά τα απόβλητα επικίνδυνα, αυτό ίσως να έχει συνέπειες και ίσως να συνεπάγεται περαιτέρω υποχρεώσεις ε, που υπέχει η Ιρλανδία βάσει οδηγία για τα ορχεία. Οπότε θα πρέπει να θεωρείται τύπου α αυτή η εγκατάσταση. Οπότε θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, σχέδια κατεπίγουσης, κατεπίγουσης ανάγκης. Περιμένουμε τις πληροφορίες που ζητήσαμε που πρόκειται να φτάσουν μέχρι τις 19 Νοεμβρίου από τους Ιρλανδούς και μετά θα κάνουμε τη δέουσα ανάλυση και θα δώσουμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που θα είναι στη διάθεσή μας στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ε, θέλουν οι συνάδελφοι να μιλήσουν. Ο συνάδελφος Μποστινάρου έχει το λόγο. Grazie, Madame Presidenta. η απάντηση που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την ε, πρόσφατη πληροφόρηση δείχνουν ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και η καταστροφή που σημειώθηκε στην περίπτωση του Μάγκερ Αλουμίνιουμ δείχνουν ε, τι κινδύνους ε, αντιμετωπίζουμε σε τέτοια ατυχήματα. Οπότε παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει όλες τις αναγκαίες ε, οικονομικές, ε, νομικές και λοιπά εγγύησεις, να μας διαβεβαιώσει δηλαδή ότι η αρχή ο Μολύνων πληρώνει, θα ισχύσει στην περίπτωση της ε, Ιρλανδίας. Ξέρετε, στην Ουγγαρία είχαν γίνει επιθεωρήσεις που λέγανε όλα πάνε πρίμα και μετά έσκασε το πράγμα. Και η Ουγγρική κυβέρνηση αναγκάστηκε να ε, επιβάλλει ένα πρόστιμο 5 δις ευρώ είναι τόσο ψηλό που δεν πρέπει να το πληρώσει. Και ούτε μπορείς να βρεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, είναι κάποια offshore εταιρεία. Δεν βρίσκεις ε, τον μολύνοντα για να εφαρμόσεις την αρχή. Ο μολύνον πληρώνει. Πρέπει λοιπόν ε, να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας, να εδρεωθεί, ούτως ώστε να μην έχουμε τα ίδια στο μέλλον, διότι η ρουμανική περίπτωση, Μπάια Μάρε, και η ουγγρική περίπτωση, Μάγκερ Αλουμίνιουμ, μας δείχνουν ότι στη θεωρία όλα πάνε πρίμα, αλλά στην πράξη δεν πάνε. Στόχος μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Να το διασφαλίσουμε αυτό. Θέλω σαφέ μήνυμα να μας δοθεί. Τι αποζημιώσεις ε, μπορεί να χρειαστεί να πληρωθούν. Όχι μόνο τι επίγοντα μέτρα θα ληφθούν, αλλά και τι χρηματικές εγγυήσεις μπορούν να υπάρξουν για να καλύψουν το κόστος μιας καταστροφής. Διότι αλλιώς, ναι μεν στα λόγια λέμε να πληρώνει ο Μολύνων, αλλά στην πράξη θα πληρώσει το κράτος. Και τώρα σε περιόδους κρίσης ε, και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, ξέρετε τι τρομερές επιπτώσεις έχουν ε, μολύνσεις τέτοιου τύπου. Συγκρίνοντας με τα προηγούμενα δύο ατυχήματα, Μπάια Μάρε και Μάγκερ Αλουμίνιου. Λοιπόν, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αναμένοντας νέα απάντηση από τις Ιρλανδικές Αρχές και μετά θα αποφασίσουμε τι θέση θα λάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι απαραίτητο να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Βέβαια, δυστυχώς πρέπει να δούμε ότι η καζόμενη επικίνδυνη ε, κατάσταση παραμένει για το περιβάλλον χωρίς λύση για έξι χρόνια. Ελπίζω οι επόμενε απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φτάσουν γρηγορότερα και αυτό να μας επιτρέψει να ενεργοποιήσουμε διαδικασίες. Αν μη τι άλλο επιβολή κυρώσεων, αλλά να απευθυνθούν σοβαρότερες προειδοποίησεις προς την Ιρλανδία, αν μη τι άλλο αυτό. Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το σημείο. Το επόμενο σημείο της μέσιας διάταξης είναι η αναφορά του σημείου 21 που προβλέπει την παρέμβαση του Αντιπροέδρου Ταγιάννη. Γι' αυτό διακόπτουμε τις εργασίες μας εν αναμονή αφήξεώς του. Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Μπορούμε να επαναλάβουμε τις εργασίες μας. Χαιρετίζω τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη. Τον ευχαριστώ που δέχτηκε να συμμετάσχει σε εργασίες της Επιτροπής μας που τροφοδοτήθηκε από τις συζητήσεις επί της αναφοράς που υπευλήθη από Ιταλό πολίτη και από άλλους υπογράφοντες για το θέμα της εγκατάστασης παραγωγής χάλιβα στον Τάραντα. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα στην Ιταλία σήμερα λόγω της ε, παρέμβασης των δικαστικών αρχών που ζήτησε, επέβαλε το να κλείσουν τμήματα της εγκατάστασης στον Τάραντα. Σε σχέση με αυτό το θέμα το Ιταλικό, από παλιά είχαν κινητοποιηθεί ενεργά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που επηρεαζόμενοι και από τις δικές μας δραστηριότητε, από τις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλαβε μέτρα προειδοποίησης κατά της Ιταλίας. Επίσης παρεπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ολοκληρώθηκαν διαδικασίες τον Μάρτιο του 2011, εκδικάστηκε η υπόθεση και το δικαστήριο καταδίκασε την Ιταλία για την δυναμία των Ιταλικών αρχών να επιβάλλουν την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε αυτό το στάδιο παραμένουν δύο εκκρεμή θέματα πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο ερωτηματικά δημιουργούνται που έχουν θέσει οι πολίτες μας, που έχουν υπογράψει το ερώτημα όσον αφορά τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το δεύτερο ερώτημα είναι ποια συγκεκριμένη δυνατότητα υπάρχει η Ιταλική κυβέρνηση να παρέμβει για υποστήριξη εγκατάσταση και με οικονομικά μέτρα που πρόσφατα υιοθετήθηκαν χωρίς να παραβιάζονται οι αρχές που απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις. Αυτά είναι τα βασικά ανοιχτά ερωτήματα για τα οποία θα παρακαλούσα να παρέμβει ο Αντιπρόεδρος ο κ. Σταγιάννη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξέρετε ότι η κατάσταση του Ήλβα στο Τάραντα είναι κάτι που δεν αφορά μόνο ένα κράτος μέλος, όχι μόνο μια σημαντική περιοχή ενός κράτους μέλους, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Βα του Τάραντα είναι το μεγαλύτερο χαλιβουργικό κέντρο της Ένωσής μας. Έχει περίπου 12.000 εργαζομένους εκεί και ας προσθέσουμε και 8.000 εργαζομένους που εργάζονται σε πανεφέρειες επιχειρήσεις. Πάρα πολλές οικογένειες λοιπόν εξαρτώνται από εκεί είναι θέμα που αφορά και τις περιβαλλοντικές πολιτικές, προστασία της υγείας των συμπολιτών μας και τις κοινωνικές πολιτικές, απασχόληση και τις βιομηχανικές πολιτικές, διότι ο χάλιβας είναι ένας, ο χαλιβουργικός τομέας είναι ένας από τους τομείς τους πολύ σημαντικούς βασικούς για την οικονομία της Ένωσής μας. Εδώ, όπως γνωρίζετε, κατ' παρελθόν συζητήθηκαν τα θέματα αυτά του ΕΛΒΑ, κατόπιν της ε, αναφοράς του κύριου Κώσιμου Φρακάσου που κατέθη το 2007 και μετά την αναφορά έγινε το 2008 έρευνα σε στενή συνεργασία με τις Ιταλικές ε, αρχές. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προκατακτικά συμπεράσματα εδώ στην Επιτροπή σας. Διαφάνει ότι η Ήλβα δεν σεβόταν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής για την πρόληψη και τον ολοκληρωμένο έλεγχο όσον αφορά τη ρήπανση. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία κατά παράβαση ε, τη, κατά της Ιταλίας. Όπως υπενθύμησε η Πρόεδρος Ματσόνη, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ανάλυση και εδώ και 1,5 χρόνο, 31 Μαρτίου του 2011, η Ιταλία καταδικάστηκε διότι δεν ε, εξασφάλισε επαρκώς το ότι όλες οι εγκατάστασεις περίπου 80 εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων και αυτή η συγκεκριμένη εγκατάσταση ε, πληρούσε τις προδιαγραφές. Εξετάζεται η από τις ε, νομικές αρχές της ε, Ιταλίας λόγω εκπομπών ρηπαντικών αρχών. Λοιπόν, στον Οκτώβριο η εισαγγελία είπε ότι οι διάφορες εγκαταστάσεις που ερευνούνται πρέπει να κλείσουν κάποιες μονάδες εγκατάστασης διότι εξέπεμπαν ρηπαντικές ουσίες και θα πρέπει μέσα σε πέντε μέρες να κλείσουν αυτά τα τμήματα ή μέχρι, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Η κατάσταση ε, φυσικά συνεχώς εξελίσσεται. Χθε η Ήλβα παρουσίασε μια πρόταση κατά, προσφυγής κατά της απόφασης και τώρα οι Ιταλικές αρχές θα πρέπει να αποφασίσουν πώς να δώσουν συνέχεια στις ε, διατάξεις εντολές που έδωσε ε, ο εισαγγελέας. Όσον αφορά τις δικές μου, τα δικά μου καθήκοντα που είμαι επίτροπος υπεύθυνο για τη βιομηχανία και σε σχέση με αυτό το γεγονός ε, λιγότερο πριν από ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα, κατόπιν πρόσκληση το πρόεδρου τη περιοχή του κ. Βέντον ε, ε, συμμετείχα στον Πάρη σε μια διάσκεψη οργανική με τον Υπουργό περιβάλλοντο Κλίνη, τον Υπουργό περιβάλλοντο, με τον Υφυπουργό ανάπτυξη τη της κυβέρνηση Δεβιτσέντη, και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Βέντολα, την τοπική αυτοδιοίκηση, εκπροσώπους της εταιρεία και εκπροσώπους ε, των διαφόρων συνδικαλιστικών δυνάμεων. Κάθε συμμετέχον δεσμεύτηκε να βρει μια λύση που θα προστατεύσει την υγεία των πολιτών και ταυτόχρονα να διαφυλάσει και τις θέσεις εργασίας. Ε, ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την υπόθεση ΙΡΒΑ. Ε, υπάρχουν τρει βασικέ ε, γραμμέ δράση που μπορούν να ακολουθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρακολούθηση. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπη παρακολουθεί τι εξελίξει στον Τάραντα και φέτο το Μάρτιο ξεκινήσαμε έρευνε μέσω του pilot του πληροφορικού συστήματο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων κοινοτικών προδιαγραφών. Η Ιταλία απάντησε στα ερωτήματα όσον αφορά την Ήλβα, επιβεβαιώνοντα ότι η εγκατάσταση του Τάραντα έχει άδεια ε, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ε, διαπιστώθηκαν ελλείψεις όσον αφορά τους διενεργηθέντες ελέγχους εντός του εργοστασίου και κυρίως όσον αφορά τις εκπομπές. Όσον αφορά το δεύτερο άξονα δράσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά πόσο γίνονται σεβαστές ευρωπαϊκοί παράμετροι για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, σύμφωνα με την οδηγία ad hoc Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2012 είχε υποχρέωση η Ιταλία να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκέντρωση ρηπαντικών ουσιών ε, βενζολίου, ε, οξυδίου του, αζότου του αζώτου και άλλων ουσιών μέχρι το τέλος του 2011 και εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να διαπιστώσει κατά πόσο ταιριάζουν οι διάφορα, τα διάφορα, οι διάφορες εκπομπές με τις προδιαγραφές. Μετά η οδηγία για την πρόληψη και ολοκληρωμένο έλεγχο της ρήπανσης. Το Φεβρουάριο φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε απόφαση που καθορίζει ε, ποια είναι η ενία της οδηγίας είναι οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες για τις εκπομπές του τομέα της χαλιβουργίας. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιούνται από τι Ιταλικέ αρχέ για να επικαιροποιήσουν την άδεια λειτουργία της εγκατάσταση του Τάραντα, την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως αποκαλείται. Ε, λοιπόν, προβλέπεται 18 Οκτωβρίου η αδειοδότηση αυτή και θα είναι το αποτέλεσμα συντονισμού κυβέρνησης, επιχείρησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επίτευξη συμφωνίας γίνεται υπό τον όρο ότι η Ήλβα θα αναλάβει την υποχρέωση να μειώσει τις βλαβερές αυτές εκπομπές και να κάνει τι αναγκαίε βελτιώσει, ούτω ώστε να ε, συμμορφωθεί με τι καλύτερε διαθέσιμε τεχνολογίε που ε, καθορίζονται και υπάρχουν το έτο 2012. Λοιπόν, ε, μέχρι το 2016 πρέπει να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τι τεχνολογίες μειώνοντας σημαντικά τα επίπεδα της ρήπανση. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου βάσει τη έρευνα που ξεκίνησε, θα πρέπει η Ιταλία να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια απάντηση όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν και να δώσει αντίγραφο τη ολοκληρωμένη αδειοδότηση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, που θα είναι επικαιροποιημένη με τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Αυτά όσον αφορά τι πτυχέ ε, τι περιβαλλοντικέ που συνδέονται με το θέμα Ήλβα Είναι θέμα που το επεξεργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τον αρμόδιο επίτροπο, ε, που είναι ο επίτροπο Ποτότσνικ. Μετά υπάρχει ένα γενικότερο θέμα που αφορά την ανταγωνιστικότητα του τομέα που όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά περνάει πολύ δύσκολες στιγμές μετά από την πτώση της ζήτησης σε όλη την Ευρώπη, την αύξηση του κόστους της ενέργειας και την αυξανόμενη πίεση από πλευράς των εξωτερικών μας ανταγωνιστών. Ε, τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του τομέα του Χάλιβα μαζί με τον Επίτροπο Άντορ ε, ξεκινήσαμε μια ομάδα εργασία που αφορά το χάλιβα, συζητά το θέμα του χάλιβα για να εντοπίσουμε τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Συμμετέχουν οι διάφορε χαλιβουργικέ εταιρείε, οι μεγαλύτερε εταιρείε, Ρίβα, το Μεντάλ κλπ. Ε, και οι κοινωνικοί εταίροι του, όλα τα συνδικάτα του, της Ευρώπης, του τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στι συνεδριάσει σαν παρατηρητής με την συμμετοχή του Προέδρου της Επιτροπής Βιομηχανίας, της κυρίας Σαρτόρη, του Πρόεδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της κυρίας Περβάνς Μπερές επίσης. Ζήτησα και το Συμβούλιο τελικά θα θέσει στην ημερήσια διάταξη του, της αυριανής συνεδριάσεως στο Λουξεμβούργο το θέμα της κρίσης της χαλιβουργίας, του Χάλιβα, Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να συζητήσουμε εν γέννη την όλη κατάσταση στον τομέα του Χάλιβα. Εκεί θα παρουσιάσω στους συναδέλφους του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας τι ακριβώς κάνουμε, κυρίως όσον αφορά την ε, βιομηχανική πολιτική. Ε, στόχος είναι να παρουσιάσουμε στο σώμα των επιτρόπων ένα σχέδιο δράσης για τον τομέα του Χάλιβα μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα Ήλβα, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ε, στις Ιταλικές αρχές, κάτι που βεβαιώνεται και από τα αποτέλεσμα μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης ε, που είχαμε με τον Υπουργό Κλίνη, που είναι Υπουργό Περιβάλλοντας της Ιταλικής Δημοκρατίας, που με επιβεβαίωσε τη βούληση της Ιταλίας να σεβαστεί και να εφαρμόσει όλες τις κοινοτικέ προδιαγραφές και διατάξεις. Ήδη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ε, εφαρμογή όλων των κοινοτικών προδιαγραφών και για την ε, διοδότηση. Όσον αφορά τα μέτρα κατά παράβαση, δεν υπάρχουν μέτρα που θα επιβληθούν στην Ιταλία σε αυτή τη φάση όσον αφορά το θέμα Ήλβα. Εμεί όμω θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την κατάσταση, λαμβάνοντα όντω υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την ποιότητα του σφαιρικού αέρα τη περιοχή του Τάραντα και τι σημαντικέ ε, αλλαγέ που υπάρχουν στον τομέα τη απασχόληση. Είμαι στη διάθεσή σα για ενδεχόμενες ερωτήσει και είμαι στη διάθεση του Κοινοβουλίου όλων των επιτροπών των αρμοδίων για να δώσω πληροφορίες που αφορούν την πολιτική μας τομέα του Χάλιβα. Να σας πω, δε, ότι αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει το έγγραφο, το σχετικό, με τη βιομηχανική πολιτική που συμπεριλαμβάνει μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλειών και δράσεις για την υποστήριξη του τομέα του Χάλιβα, που θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδης για την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό στα πλαίσια του σεβασμού των διάφορων περιβαλλοντικών προδιαγραφών και των στόχων 2020-2020. Ε, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ εσάς και ευχαριστώ και την Πρόεδρο για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Ταγιάννη. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Ο κύριος Γιάρ ζήτησε το λόγο. Με συγχωρείτε, δεν είχα στήσει το λόγο. Μετά, μετά, μετά, μετά μπορεί. Α, ευχαριστώ. Ριβελίνη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο Ταγιάννη για τα δύο θέματα στα οποία έδωσα απαντήσει σήμερα. Νομίζω ότι μεγάλη προσοχή δίδεται στην Ιταλία τα θέματα αυτά, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά το θέμα της ανταγωνιστικότητας του τομέα, Περιμένουμε τη συνεδρίαση που ανήγγειλε ο, Επίτρο, ο Επίτροπος Ταγιάννη ε, διότι στην αντιπροσωπεία Ευρώπης-Κίνας επανειλημμένα συζητήσαμε τον ανταγωνισμό σαν προϊόν που είναι ουσιαστικό προϊόν, θεμελιώδες προϊόν. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της συνεδριάσεως για να μπορέσουμε να συζητήσουμε εκ νέου ενδεχομένως το θέμα με τους ε, Κινέζους ομολόγους μας. Όσον αφορά το θέμα Ήλβα, πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε προσεκτική αξιολόγηση των όσων συνέβησαν, κύριε Επίτροπε. Ε, διότι, όπως είπε και η εισαγγελία, είναι η έλλειψη επενδύσεων που οδήγησε στην καταστροφή ε, του Τάραντα. Εγώ θα ήθελα να επιθυμίσω στους συναδέλφους ότι το κράτος παρήγαγε ε, και στο, στο, στο Ντάραντα και στο Χάλιβα, διότι ήταν κρατική επιχείρηση. Τον Ιούνιο ε, πήγα κοντά στον Πέργαμο στην κατάσταση και πάντα στη Βόρεια Ιταλία παρήγαγε με σωστό τρόπο σε αυτή την εγκατάσταση το προϊόν. Δεν ρηπαίνει το περιβάλλον και δεν υπονομεύεται η υγεία των εργατών και των εργαζομένων. Στον Πανιόλι και στον Τάραντα το κράτος παρήγαγε ε, ε, μολύνοντας τους εργαζομένους και καταστρέφοντας το περιβάλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Μετά σχεδόν δωρεάν ε, έδωσε την επιχείρηση στους ιδιώτες χωρίς να είναι σίγουρο το κράτος ότι γινόταν οι ε, σωστές επενδύσεις να προστατεύεται η, περιοχή. Και σαν Ευρωπαίος ε, πολίτης ρωτώ, τι διαφορά έχει αυτή η τραγωδία με αυτό που έγινε στο Σεβέζο, στο Σοβέζο, ε, όπου εκεί οι Ελβετοί ήθελαν πιο στα νότια να παράγουν για να αποφύγουν προβλήματα και συνέβη αυτό που συνέβη. Ή στην Ινδία, όταν συνέβησαν αυτά τα τραγικά γεγονότα που θυμούνται όλοι. Το Ιταλικό κράτος θα πρέπει να παρέμβει και θα πρέπει να παρέμβει το ταχύτερο δυνατόν για να αποκατασταθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος, να εξασφαλιστεί στους εργαζομένους δουλειά και να αποφευθεί μια συνέχιση αυτής της προφανούς αδικίας και ντροπή. Περιμένω μετά η Ευρώπη και το λέω σαν Ιταλός Ευρωβουλευτής. Περιμένω η Ευρώπη να παρέμβει με τον πιο σωστό και σκληρό τρόπο. Να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Ιταλία που είναι υπεύθυνη για όλα αυτά να διαπιστωθεί γιατί στη Βόρεια Ιταλία πάντα γινόταν η παραγωγή του ίδιου προϊόντος του χάλιβα χωρίς να, να ρηπαίνονται, να μολύνονται οι πάλι και να σφαγιάζονται οι πάλι κάτι που συνέβη στον, στην Νότια Ιταλία, στο Τάραντο και στο Πανιόλι. Και μετά, την απάντησή σας, έστειλα επιστολή και σε εσάς και στα, στην Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Λουξεμβούργο ε, ζήτησα για τους υπαλλήλου εκείνους, για τους εργαζόμενους που εντωμεταξύ μεταξύ ε, είναι στην ανεργία ε, από, την κατάσταση, από τη μονάδα Ήλβα ε, να πάρουν χρήματα από το Ταμείο της Παγκοσμιοποίηση που έχει 500 εκατομμύρια ευρώ αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης ενεργοποιήθηκε πλέση για 7 υποθέσεις στην Ιταλία μόνο μία ενεκρίθη εδώ θα έπρεπε να γίνει. Είναι μια πρόταση δική μου να χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό, να ενεργοποιηθεί αυτό το ταμείο για αυτούς τους ανθρώπους. Και εδώ κλείνω, ε, Πρόεδρε Ματσόνη και Επίτροπε Ταγιάννη. Εδώ στην Ευρώπη συζητούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών του κόσμου. Ινδιά, Ινδών, Κινέζων, Αφρικανών και είναι Και θα πρέπει να πολεμήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ε, πολιτών και για τους εργάτες της Νότιας Ιταλίας που με ψήφισαν. Δεν πρέπει να μιλήσω, να συζητήσω για τα δικαιώματά τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα εκείνων που με ψήφισαν. Ε, λέμε στην Ιταλία κάτι επίκαιρο. Αυτό που είναι καλό να κάνεις για σένα, καλό να κάνεις και για, και για τους άλλους. Αυτό θέλω να πω. Και σε ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ, κύριε Ριβελίνη. Ζανώνε. Ο κύριο Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ διαρωτώ με, όσον αφορά το θέμα Ήλβα, μήπως είναι η κορυφή του παγόβουν αυτή και διαρωτώ με πώς ένα θέμα τόσο σημαντικό που βασίζεται στα Ιταλικά ε, χρονικά και τα Ευρωπαϊκά πώς ετέθη στο φως μόνο ε, χάρη στην ε, εισαγγελία. Η έλεγχη του κράτους μέλους, σε αυτή την περίπτωση της Ιταλίας, όσον αφορά το σεβασμό των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, ήταν επαρκής, υπάρχουν και διαρωτώμε Και κάτι άλλο που διαρωτώμε Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει καλύτερο σύστημα που θα ενεργοποιούσε ούτω ώστε αυτοί οι κανόνες, οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας να γίνονται σεβαστοί μέσω ελέγχου περιοδικού ενδεχομένως με την αποστολή επιθεωρητών σε διάφορα κράτη-μέλη. Ε, να υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη παρουσία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ε, πολύ σημαντικό θέμα. Μας λένε ίσως ότι οι έλεγχοι δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν δεν λειτουργούν. Πόσες υποθέσεις ή τύπου Ήλβα υπάρχουν στην Ιταλία που δεν γνωρίζουμε και δεν γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύουμε το περιβάλλον και πάνω απ' όλα την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν άλλε υποθέσει. Υπάρχουν χαλιβουργία, άλλε χαλιβουργίε. Σε όλη την Ευρώπη και την Ιταλία υπάρχουν εγκαταστάσει ε, που μπορούν να κάψουν τα πάντα εκεί. Και τα απόβλητα πηγαίνουν μετά στα απόβλητα και μπαίνουν σε διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται και στι οικοδομέ. Υπάρχουν εκατοντάδε καυστήρε. Η, Ένωση Γιατροί για το Περιβάλλον έκανε μια εκστρατεία που μιλά για το μητρικό γάλα, με αυτό εννοώ ε, γάλα των μητέρων, μητρικό γάλα. Διότι κάποτε δεν έχει μεταφραστεί σωστά αυτά. Μητρικό γάλα λοιπόν που έχει μολυνθεί από διοξίνη. Υπάρχουν δεκάδε περιπτώσει στην Ιταλία που μετά από ανάλυση του μητρικού γάλακτο ανακαλύπτεται ότι υπάρχει διοξίνη ε, στο, στην πρώτη τροφή που θα έπρεπε να είναι η πρώτη τροφή των ε, παιδιών, των μωρών. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Ευρώπη, η Ιταλία, όλοι να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε ένα σύστημα ελέγχου όσον αφορά το μητρικό γάλα, παραδείγματο χάρη. Διότι έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δεκάδε, εκατοντάδε μάλλον υποθέσει ήλβα, τύπου ήλβα, που ακόμα είναι άγνωστε σε εμά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, χάρη στην, ε, στην εισαγγελία ξέρουμε τι έγινε εδώ. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθορίσει αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις και μολυσμένο, το μολυσμένο μυτικό γάλα με διοξίνη μας το δείχνει αυτό. Ε, ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Τζανόνε. Ο κύριος Γιάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Αν κοιτάξει κανείς την ε, Επιτροπή, δύο πράγματα προκύπτουν αμέσως. Το πρώτο είναι ότι λειτουργεί η διαδικασία. Διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή αντέδρασε, της κάλεσε την Ιταλία να τηρήσει ε, τις ε, διατάξεις και εφόσον αυτό δεν έγινε υπήρξε προσφυγή. Αυτές είναι οι καλές ειδήσεις θα έλεγα. Αλλά Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι δεν είναι δυνατόν κάθε κράτος μέλος να επιχειρεί να ελέγξει κάθε επιχείρηση. Βεβαίως έχει και η Επιτροπή την υποχρέωση να την πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που με απασχολεί εμένα και το ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι είναι είναι ότι δεν ήταν λεπτομέρειες ε, οι παραβιάσεις, αλλά ήταν ιδιαίτερα βλαβερές οι ε, χημικές ουσίες που εκλείονταν στο περιβάλλον, πόσο πολύ κράτησε η διαδικασία μετά από αυτό. Είναι ουσίες που μπορούν να ε, κάνουν ζημιά στην υγεία των πολιτών. Έπρεπε λοιπόν να έχουν αντιμετωπιστεί νωρίτερα διότι μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τελικά οι μολύνοντες κάνουν καθυστέρηση. Η όλη διαδικασία κρατάει πάρα πολύ. Χαίρομαι λοιπόν που λειτουργήσε η διαδικασία. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι δεν θα συνέβαιναν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη. Καλά, αυτό το περιμένουμε ακόμη. Αλλά θα μπορούσαμε εμεί να περιμένουμε ότι όταν υπάρχουν τόσο σοβαρέ για την υγεία επιπτώσει από τι παραβιάσει, τότε θα έπρεπε να υπάρχει ταχύτερη αντίδραση. Το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με τι τεχνολογίε. Δεν υπάρχει μόνο ένας παραγωγός. Υπάρχουν άλλοι παραγωγοί που ε, αντιμετωπίζουν καλύτερα τις διαδικασίες αυτές. Για μένα το θέμα είναι πώς θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία προς το συμφέρον των αναφερόντων, προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτόρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ και για τη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σήμερα στην Επιτροπή μας πάνω σε αυτό το θέμα που σωστά λόγω της κατάστασης που διαπιστώνουμε γίνεται κεντρικό θέμα της συζήτησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το άλλο άρρηκτα συνδεδεμένο θέμα, την οικονομική κρίση και το τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση και να βγούμε από την κρίση. Και εγώ σήμερα το πρωί στη συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Βιομηχανίας συζήτησα μαζί τους και αξιολόγησα την παρουσίαση ερώτησης για διεξαγωγή συζήτηση στην Ολομέλεια με θέμα ακριβώς τη χαλιβουργία τον τομέα αυτό. Η συζήτηση δεν μας επέτρεψε να εισαχθεί το θέμα αυτό ήδη στην επόμενη μυρίσια διάταξη της επόμενης ε, Ολομέλειας. Όλοι οι συντονιστές, όλες οι παρούσες ομάδες συμφώνησαν στη Σύνοδο του Νοεμβρίου να συζητηθεί το ζήτημα. Ε, θα προταθεί από την Επιτροπή Βιομηχανίας. Για να πω ότι τώρα πια σωστά η προσοχή έχει επικεντρωθεί. Όπως σωστά το έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ένα θέμα που το παρατηρούν όλοι στην Επιτροπή Βιομηχανίας διότι είναι ένα θέμα που συνδέεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και μπορούμε να την υπερασπιστούμε και στα πλαίσια εσωτερικής και πώς έχουμε δυνατότητα εντός κρατών μελών να αυξήσουμε, να υποστηρίξουμε και να βελτιώσουμε τη βιομηχανία μας και σε σχέση με τις πολιτικές που έχουμε εντός κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις τρίτες αγορές, τις αγορές τρίτων χωρών. Είναι δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι δικό μας εσωτερικό, η διαφύλαξη, η προφύλαξη και επαναπροώθηση βιομηχανία και δεύτερο σημείο, οι σχέσεις με άλλες χώρες του κόσμου για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς να αντιμετωπίσουμε σωστά το ζήτημα του ανταγωνισμού και της παραγωγικότητας εναντί αυτών των χωρών. Σίγουρα τα επεισόδια αυτά που συνέβησαν αυτούς τους μήνες και η αναφορά που υπευλήθη καταδεικνύουν το πώς χρειάζεται να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Όπως και αυτά που συζητήσαμε το πρωί. Το θέμα Ήλβα του Τάραντα. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Από τη μία πλευρά τη διαφύλαξη της βιομηχανίας μας, ε, προστασία της απασχόλησης, θέσεων εργασίας, προστασία και υποστήριξη ανάπτυξη οικονομίας. Από την άλλη πλευρά κάτι εξίσου σημαντικό, πιο σημαντικό, πρέπει να εγγυηθούμε τη ισχύουσα νομοθεσία με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα τα οποία έχουμε σήμερα επιτάπητος μπροστά μας. Όπως υπογράμμισαν πολλοί συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πιθανότατα και το ένα και το άλλο θα πρέπει να ειδωθούν σε δύο πλαίσια, εθνικό και ευρωπαϊκό. Να μην γίνει άλλο ένα στοιχείο που θα διαφοροποιεί τις πολιτικές μιας χώρας εναντί μιας άλλης. Θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ότι οι παραγωγικές μονάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σέβονται τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και εγγυώνται την υγεία εκείνων που εργάζονται εκεί και των πολιτών που κατοικούν κοντά σε αυτές τις μονάδες και από την άλλη πρέπει να έχουμε μια πολιτική που θα υπερασπίζεται απόλυτα τις θέσεις εργασίας, την απασχόληση και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε μπροστά μας. Μπορούμε να προχωρήσουμε όμως μαζί, πρέπει να προχωρήσουμε μαζί, είναι μια μεγάλη αποστολή που ανατίθεται και σε αυτό το επίπεδο, ξέρω, σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά με μεγάλη προσοχή πλευράς του Κοινοβουλίου που θα παρακολουθήσει την όλη διαδρομή. Το το συζητήσαμε εδώ σήμερα το πρωί δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα που συζητείτε, πόσο σημαντικές είναι οι συζητήσεις και πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτά τα δύο ζητήματα τα οποία θα πρέπει από κοινού να εξεταστούν σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Μετά μπορούμε να θέσουμε και το στόχο να πούμε ότι όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη θα πρέπει να ε, παράγονται με σεβασμό των ε, δικό μας, της δικής μας νομοθεσίας αυτών των προδιαγραφών. Ξέρω ότι αυτό είναι καυτό ζήτημα. Όπως το κάναμε με τριοπαθώς άλλους τομείς, στον υπόλοιπο κόσμο θεωρητικά ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμω μπορούμε να πούμε ότι τα προϊόντα τα οποία εισάγονται και διαθήκονται στο εμπόριο στην επικράτειά μα θα πρέπει να παράγονται με πλήρη σεβασμό των προδιαγραφών που ε, θέτουν και το πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Σαρτόρη, λέει η Πρόεδρο. Ο κ. Μποστινάρου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ταγιάννη για την συμμετοχή του. Θα μιλήσω τώρα ρουμανικά, αν μου επιτρέπετε. Είμαστε αδελφοί σε κάθε έννοια. Λοιπόν, συζητούμε εδώ ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα δραματικό θα έλεγα πρόβλημα Και ουσιαστικά φταίνε και τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν, όχι μόνο η Ιταλία. Το λέω αυτό γιατί έτσι κατέστη ε, δυνατή παραβίαση ευρωπαϊκής οδηγίας με πολύ συστηματικό τρόπο και επίμονο τρόπο. και υπήρχε η ουτοπία ότι κάτι θα γίνει τελικά και κάτι θα, κάπως θα διορθωθεί η κατάσταση. Εδώ όμως μιλάμε για την εξέβρεση λύσης για μια πάρα πολύ σημαντική περίπτωση ρήπανσης εν μέσω μία σοβαρής κρίσης. Μεγάλης κρίσης η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ε, τη δουλειά τους και να μην έχουν ελπίδα να βρουν μια άλλη. Οι ελπίδες τους δε ότι θα τους βοηθήσουμε εμείς από εδώ όλο και μειώνονται. Η περίπτωση Ήλβα επιβεβαιώνει αν αυτό χρειαζόταν ε, ότι άλλη μία τέτοια αυταπάτη, άλλη μία το οποία πέθανε. Το κράτος ήθεσε να λέμε ότι πάντα φταίει και οι ιδιωτικοί φορείς, οι ιδιωτικοί παράγοντες ως εκτάβματος ε, θα σώσουν την κατάσταση. Η περίπτωση Ήλβα όμως επιβεβαιώνει ότι η ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιριών δεν βελτίωσε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, επιδόσεις. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στην Ιταλία, αλλά και σε άλλα μέρη. Σκεφτείτε την κλίμακα των ιδιωτικοποιήσεων στη Ρουμανία, για παράδειγμα. Οι εν λόγω ιδιωτικοποιήσεις οδήγησαν σε κλείσιμο και καθάριση, ε, πτώχευση ολόκληρων τομέων, ολόκληρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Με την περίπτωση Ήλβα σήμερα αλλά και με άλλες τέτοιες υποθέσεις βλέπουμε, διαπιστώνουμε την απουσία μιας πραγματικής ε, βιομηχανικής στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας παγκόσμιος οικονομικός παράγοντας παρόλα αυτά. Έχουν εκπονηθεί εθνικές στρατηγικές, οι οποίες όμως είναι ανταγωνιστικές μία προς την άλλη. Δεν υπάρχει όμως μια ευρωπαϊκή στρατηγική ώστε να σώσουμε πραγματικά σημαντικού για την Ευρώπη τομεί οικονομική δραστηριότητα. Χαίρομαι πολύ που άκουσα σήμερα τον Επιτρόπο Ταγιάννη να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλου αποφάσισε να αναπτύξει μια τέτοια στρατηγική. Θα ήθελα να το πιστέψω. Θα ήθελα να γίνει πραγματικότητα αυτή η στρατηγική, να είναι μια πλήρης στρατηγική που θα καλύπτει όλο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη, τα 27 και τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Υπάρχουν κλάδη, βιομηχανική σε πολλές χώρες, σε πολλά μέρη που πλήττονται, πλήττονται πολύ σοβαρά. Ίσως να μην είναι η ρήπανση τόσο σημαντική όσο στην περίπτωση, αλλά υπάρχουν τέτοια προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Πριν ολοκληρώσω την παρεμβασή μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε κάτι κύριε Πίτρο. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αναφέρονται τα δικαιώματα και υποχρεώσει και των Ευρωπαίων εισαγωγέων, που είναι πολίτε και αυτοί. Είναι βέβαια πρόσωπα νομικού δικαίου, νομικά πρόσωπα. Θα πρέπει όμω και αυτοί να έχουν ε, τα ίδια δικαιώματα και τι ίδιε υποχρεώσει. Προ όφελο τη διαφύλαξη περιφρούρηση αυτών των βιομηχανικών τομέων τη Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενδώσουμε σε εμπορικά και βιομηχανικά λόμπι σε βάρο άλλων χωρών. Γιατί όσοι εισάγουν παράδειγμα χάρη χάλιβα από την Κίνα, είναι μεγάλοι Ευρωπαίοι. Είναι Ευρωπαίοι πρωταγωνιστέ. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει όμω ε, να επιφυλάσσει ισότιμη μεταχείριση προ όλου. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για μια χαλιβουργία που θα διατηρήσει, θα διατηρηθεί ζωντανή στην Ευρώπη. Αλλιώ μπορούμε να κάνουμε την κηδεία τη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Er Θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Παρόλο που δεν σχετίζεται η γλώσσα μου με τα ρουμανικά ή τα ιταλικά. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος, ε, ανέφερε τις μεγάλες δυσχέρειες που έχουμε ε, σε πολλές χώρες ε, όσον αφορά τη χαλιβουργία. Στη Δανία παλιότερα είχαμε ε, μεγάλη παραγωγή χάλιβα ενώ τώρα υπάρχει μεγάλη ενεργή σε αυτό το τομέα. Και για να αποφύγουμε λοιπόν ενεργή σε αυτό το τομέα μας πιέζουν να αποδεχθούμε μειωμένες περιβαλλοντικές διατάξεις και το τελικό αποτέλεσμα στην ε, Δανία ήταν ε, να καταργηθεί η χαλιβουργία. Δεν είναι σωστό. να προσπαθούμε να εξαιρεθεί η βιομηχανία μας από τις ε, απαιτήσεις και τις διατάξεις. Ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε και να κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία μας είναι μόνο εάν ανταποκρινόμεθα στις υψηλότερες περιβαλλοντικές διατάξεις ε, και άλλες διατάξεις, ούτως ώστε να είμαστε πρωτοπόροι. Και τα προβλήματα μόλυνσης από την ε, χαλιβουργία είναι πολύ σοβαρά, όπως διαπιστώνουμε και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ε, είναι προς όφελος κανενός να κάνουμε περιβαλλοντικές παραχωρήσεις. Στην ουσία περνάμε τα προβλήματα στο μέλλον. Όλοι γνωρίζουμε τι ισχυρές ε, πιέσεις και τι λόμπι υπάρχουν ε, και έρχονται και σε εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητούν μείωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Αλλά η στρατηγική αυτή σημαίνει ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού θα, δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν με αυτή την πολιτική υπερπροστατευτισμού τις άλλες βιομηχανίες σε άλλα μέρη του κόσμου. Σας ευχαριστώ λοιπόν που απαιτείτε να τηρούνται οι αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Μην ξεχνάτε ότι η χαλιβουργία παίζει μεγάλο ρόλο και για την ανακύκλωση. Ένα μεγάλο τμήμα των εγκαταστάσεων ε, των χαλιβουργίων μας ε, λαμβάνουν ως πρώτη ύλη ε, ήδη χρησιμοποιημένα προϊόντα χάλιβα ε, και τα ανακυκλώνουν. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να γίνονται παράλληλα με την ε, τήρηση των διατάξεων για την υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ να μείνει ανοιχτή παρακαλώ αυτή η αναφορά. ευχαριστώ. Να μείνει ανοιχτή αναφορά, συγγνώμη. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω σε αυτά που θα πω τα όσα είπαν οι συνάδελφοί μου Ιταλοί, αλλά και οι εκπρόσωποι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην παρέμβασή μου ε, θα ήθελα να είμαι μια φωνή που ενώνεται με τη φωνή των άλλων συναδέλφων. Πάνω απ' όλα ευχαριστώντας σας που είσαστε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ Επίτροπε Ταγιάννη που αποφασίσατε να έρθετε εδώ μαζί μας σήμερα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα όπως είναι αυτό της μεγάλης βιομηχανίας που πάντα ασχολείται με αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίω αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή των δυσκολιών των οικονομικών για όλα τα κράτη-μέλη, ε, είναι σημαντικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται και για θέματα ευαίσθητα όπως είναι το περιβάλλον, τα κοινωνικά ζητήματα. Λοιπόν, θέλω η φωνή μου να ενωθεί με εκείνη των συναδέλφων που πήραν το λόγο για να υπογραμμίσω το πόσο επίκαιρο είναι τώρα που πρέπει να πλησιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πολίτες που έχουν μείνει πίσω. Διότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 και στον προπολογισμό του 2013 που εγκρίναμε πρόσφατα στην Επιτροπή Προπολογισμών του Κοινοβουλίου έγινε λόγος μόνο και αποκλειστικά για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και είναι σωστό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ανάπτυξη και για ανταγωνιστικότητα αλλά δεν θα πρέπει να λησμονούμε να ξεχάσουμε και εκείνους που δυστυχώς θα μείνουν πίσω. Δεν θέλουμε αυτοί οι Ευρωπαίοι πολίτες να μείνουν πίσω. Λοιπόν, θα σκεφτούμε, α θυμηθούμε τους εργάτες της Σίλβα, του Τάραντα, κυρίως σας δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε κοντά σας. Υπενθύμησε ο κ. Ριβελίνη το Ευρωπαϊκό Ταμείο για ε, την παγκοσμιοποίηση ε, είχαμε θεσπίσει, ε, το συζητούμε στο Κοινοβούλιο τελευταία δυόμιση χρόνια, να ζητώ να υποστηρίξετε την ενεργοποίηση αυτού του ταμείου για να υποστηριχθούν Ευρωπαίοι πολίτε. Σήμερα μιλάμε για την Ήλβα, για τον Τάραντα. Αύριο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια άλλη Ήλβα που υπάρχει, παραδείγματο χάρη στη Ρουμανία, που θα μπορούσε να υπάρχει στη Δανία. Σήμερα μιλάμε για αυτή την Ιταλική υπόθεση, αύριο για ρουμανικό θέμα και έτσι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Ε, Γιάρο, κύριος Γιάρο. Κυρία Πρόεδρε, συμπληρώνοντας αυτά που είπαν η Ματέρα και ο Όκεν, πρώτα απ' όλα να προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Οι προηγούμενοι είπαν σωστά και τόνισαν ότι βεβαίως έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο η αναφορά, αλλά η ουσία της ε, είναι πολύ ευρύτερη Ίσως σε συνδυασμό με την ε, Ήτρε να ήταν σκόπιμο να επιχειρήσουμε να υπάρξει ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια για να μπορέσει να συζητηθεί το θέμα αυτό και στην Ολομέλεια γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό επειδή λοιπόν έχει πολύ ευρία πύχηση το θέμα αυτό δεν θα μου αρκούσε απλώς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά Παρακαλώ λοιπόν να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια ω ψήφισμα. Έχουμε δικαίωμα ω Επιτροπή Αναφορών, εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κύριος Μπορκέτσιο, και μετά θα δώσουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο. Κύριος Μπορκέτσιο, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ενώνω τη φωνή μου και με τους άλλους που ευχαριστήσαν καταρχάς τον Επίτροπο για την παρουσία του και για το ρόλο που παίζει ο αντιπρόεδρος του Κουσταγιάννη Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κόζημο Φρακάσο, αυτό τον κύριο από το 2007 πολεμά και στράφει προς την Ευρώπη. Διότι φαντάζομαι ότι πρώτα θα στράφει προς την τοπική, τοπικές δικαστικές αρχές και το 2012 διαπιστώθηκε, διαπίστωσε η δικαστική αρχή ότι πεθαίνω τον καρκίνο ανθρωπική. Θα μπορούσαν να διαφερθούν και άλλε χώρες για την, για την έρευνα, για το ερωτηματικό που θα θέσουμε όλοι. Πόσοι παρόντες ιδιοκτήτες τη ΣΥΛΒΑ δέχτηκαν να αγοράσουν από το κράτος αυτό το τεράστιο ερείπιο με τα τεράστια προβλήματα που δεν επηρεούν τις προδιαγραφές. Διότι ε, ισχύσαν αυτά που ισχύουν στην Ιταλία και στην Νότια Ιταλία διατηρούνται στη ζωή βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα μη πληρώντας περιγραφές των ε, πολιτισμένων χωρών ούτε τους εργαζόμενους και τους πολίτες της ε, περιοχής γιατί εγγυούνται απασχόληση συμφωνούν με τις διάφορες ε, συμφωνίες. δεν είναι μόνο θέμα μιας χώρας που δεν ασχολείται με την υγεία των πολιτών, είναι θέμα βιομηχανικής πολιτικής. Όλες αυτές οι βιομηχανίες που δεν παράγουν επαρκώς και για τις οποίες δαπανώνται πολλά χρήματα, είναι μια σιδερένια μπάλα στο πόδι της Ευρώπης που δεν μπορεί να αναπτυχθεί βιομηχανικά, γιατί σέρνει αυτή τη μεγάλη σιδερένια μπάλα. Προτείνω στον πρόεδρο Ταγιάννη να το λάβει αυτό υπόψη όταν θα πολεμήσει, που ξέρει πολύ καλά πώς πολεμάει στα ευρωπαϊκά βήματα για να δώσει τη μεγάλη μάχη της ανταγωνιστικότητας. Συμφωνώ απόλυτα με τις ευφυείς και ισορροπημένες θέσεις που εξέφρασε η Πρόεδρος η κυρία Σαρτόρη. Δεν θα πρέπει να ε, κρατάμε σε ζωή σαρκοφάγους μη παραγωγικούς, παραγωγικές. Θα πρέπει να ακολουθηθούν άλλα μοντέλα ανάπτυξης περιοχές αυτές. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και κυρίως των, όπως των πολιτών της Νότιας Ιταλίας όπως του Κόσμου Φρακάσο δεν θα πρέπει να τους αφήνουμε να ξεγελιώνται από κακές πολιτικές που εφαρμόζονται. Ευχαριστώ κύριε Μποργέσου, ευχαριστώ όλους. Δίνω εκ νέου το λόγο στον Αντιπρόεδρο τον κύριο Ταγιάννη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάνω από όλα που ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση επί ενός θέματος που είναι τόσο σημαντικό εντός αυτής της επιτροπής στην οποία συμμετείχα από το 1994 μέχρι το 1999. Οπότε είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που επιστρέφω ανάμεσά σας υπό την ιδιότητα του Επιτρόπου διότι είναι η Επιτροπή που είναι πιο κοντά στους πολίτες, διότι άμεσα χωρίς άλλα φίλτρα δέχεται άμεσα τις ανησυχίες. Ακούει τις ανησυχίες των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ξεκινούσα από την παρατήρηση της κυρίας Σαρτόρη και του κυρίου Γιάρ ε, Μποστινάρου και του κυρίου Μποργέτσιο. Στις ε, παρεμβάσεις τους έθεσαν το γενικότερο πρόβλημα, το γενικό πρόβλημα, δηλαδή σχέση μεταξύ βιομηχανικής πολιτικής και περιβαλλοντικής. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένο και το είπα και κατά τη διάρκεια τη ακρόασή μου όταν ήμουν υποψήφιος επίτροπο για τη βιομηχανία. Είναι ένα γάμος που μπορεί να διοργανωθεί μεταξύ ε, περιβαλλοντική πολιτική και βιομηχανική πολιτική. Ίσως θα είναι ένα γάμος συμφερόντων, όπως λεγόταν κάποτε, αλλά καμιά φορά αυτοί οι γάμοι συμφέροντος ε, τα πηγαίνουν καλύτερα από τους γάμους από έρωτα. Ε, το έγγραφο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει αύριο όσον αφορά τη νέα βιομηχανική πολιτική εδράζεται ακριβώς επ' αυτής της υποθέσεως. Στόχος μου είναι σαν αντιπρόεδρος, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφήσω στο τέλος της πενταετίας ένα σαφέστατο μήνυμα. Η Ευρώπη επέστρεψε στην νέα βιομηχανοποίησή της. Ε, να αναβιομηχανοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι βιομηχανοποιήθηκε κατά το παρελθόν. Η βιομηχανία που συζητούμε σήμερα δεν είναι η βιομηχανία του 1980, δεν είναι του 1990. Θα πρέπει να είναι βιομηχανία ποιοτική, μια βιομηχανία που βασίζεται επί της green economy, επί των οικολογικά συμβατικών ε, συστημάτων και το στατηγικό έγγραφο που θα εγκρίνουμε αύριο, ακριβώς αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί στόχος που θέτουμε είναι να επιστρέψουμε σε μια βιομηχανία που θα είναι το 20% του ΑΕΠ. Σήμερα ξέρετε ότι είμαστε κάτω από το 17, περίπου 16,6%. Ε, θέλουμε στα 3,20 που έχουμε στόχους στους κοινοτικούς να βάλουμε και ένα τέταρτο 20 που θα είναι αυτό που θα συνδέεται με την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Σας λέω σύντομα ποια είναι τα θέματα επί των οποίων βασιζόμαστε. Δεν σας διανέμω το κείμενο όμως για λόγους ε, σωστής αντιμετώπισης του σώματος γιατί θα εγκριθεί ένα γράφω αύριο. Σας λέω όμως τι θέλουμε να επεξεργαστούμε, πώς θέλουμε να κινηθούμε. Θέλουμε να βασιστούμε επί κάποιων οριζοντίων κριτηρίων ε, ούτως ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής που θα βασίζεται επί κάποιων αξώνων βασικών όπως πρόσβαση στην πίστοση που είναι βασικότατο θέμα για τις επιχειρήσεις που θα βασίζεται στην ανάπτυξη της εσωτερική αγορά, θα βασίζεται επί της καινοτομίας και της έρευνας που είναι θεμελιώδη μέσα για να είμαστε ανταγωνιστικοί, έρευνα και καινοτομία που θα εφαρμόζονται όλο και περισσότερο στην βιομηχανική πολιτική. Θα βασιζόμαστε επίσης επί κάποιων θεμελιωδών ζητημάτων που μετά έχουν και συνέπειες στο σύνολο της βιομηχανίας της ε, κατασκευαστικής και μη green economy, πράσινη economy, βασικές τεχνολογίες και enabling technologies, το μέσο του διαστήματος, ο τομέας των οικοδομών που οι οικοδομές θα είναι συμβατές με, τα, με τις οικολογικές προδιαγραφές. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η ανακοίνωση είναι καρπός 2,5 ετών εργασιών. Όπως γνωρίζετε παρουσιάσαμε στις αρχές της περίοδου Μπαρόζο 2 ένα έγγραφο για τη βιομηχανική πολιτική, μία για την πολιτική της καινοτομίας, εδώ και μερικού μήνε διοργάνωσαμε τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεγάλη εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, παρουσία του Τζέρεμι Ρίφκιν για να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική που θα είναι πραγματικά green, πραγματικά πράσινη, που θα επιτρέπει και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των οχημάτων, όχι μόνο το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχω υπόψη μου όταν το λέω αυτό, αλλά την ε, ανάπτυξη υποδομών που συνδέονται με τις μεταφορές με σιδηροδρόμους, ε, η στρατηγική για τα ναυπηγεία για να έχουμε όλο και πιο πράσινα πλοία και που ρηπαίνουν λιγότερα τα πλοία μας. Θα πούμε και στα κράτη-μέλη πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα, πώς θα μπορούν να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα ευρωπαϊκά ταμεία από τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να έχουμε αυτού του είδους την πολιτική για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Βεβαίως η ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς είναι θεμελιώδης σημασίας. Φυσικά ή μάλλον να το πω καλύτερα τις προάλλες το Συμβούλιο ενέκρινε οριστικά ένα κείμενο που ενέκρινε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' προτάσεώς μου για την τυποποίηση που είναι η πρώτη νομοθετική πράξη του Internal Market Act 1 και αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ευρύτερο της βιομηχανικής πολιτικής που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και περιβαλλοντικές πτυχές, διότι το κόστος της ενέργειας είναι κάτι σημαντικό. Και γι' αυτό εξακολουθούμε να εργαζόμαστε και για την εξοικονόμηση ενέργειας, που δεν πρέπει να υποτιμάται. Γι' αυτό μιλώ για τη βιομηχανία των οικοδομών που θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές. Και όλο το πρόβλημα συνδέεται με τις πρώτες ύλες και το λέω αυτό για αυτούς που είναι πιο ευαίσθητοι όχι μόνο για τη βιομηχανική πολιτική, αλλά και την περιβαλλοντική πτυχή, ότι θα ξεκινήσει το Innovation Partnership που αφορά την ανακύκλωση, την υποκατάσταση και την εξαγωγή των πρώτων υλών. Λοιπόν, και το θέμα των πρώτων υλών θα αποτελεί ένα κομμάτι αυτή τη στρατηγική. Κανένα τομέα δεν θα αποκλείεται, θα εξαιρείται. Μιλάμε μια στρατηγική. Είναι ένα σφαιρικό όραμα ε, τη βιομηχανική πολιτική που είναι καρπό 2,5 ετών εργασιών και επαναλαμβάνω, θα ήθελα να αφήσω σαν σημάδι της παρουσίας μου οι πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δουλειά που υπενθύμησε και ο πρόεδρος Μπαρόσο όταν σας μίλησε για την κατάσταση στην Ένωση, να δείξω ότι είναι η βιομηχανική πολιτική θεμελιώδη σημασία να ξεπεραστεί η κρίση και να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Εντό τη πολιτική βιομηχανική υπάρχει και η πολιτική του Χάλιβα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει σεβαστού του νόμου, να γίνουν σεβαστοί οι νόμοι. Ήδη υπάρχουν οι κανόνε και είναι αρκετά αυστηροί, όπω υπενθύμησα και στην εισαγωγή μου και όπω υπενθύμησε πολύ σωστά η Πρόεδρο Ματσόνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα θέματα που συζητούμε σήμερα, και συγκεκριμένα, παρενεύει. Έγινε διαδικασία παράβασης, παραβίασης που εκκρεμεί Είχαμε απόφαση της... Ε, ξεκίνησε μάλλον αυτή η διαδικασία και έχουμε απόφαση του δικαστηρίου. Υπάρχει αυτή η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν έχει όμως μέσα αστυνομικού χαρακτήρα στη διάθεσή της. Υπάρχουν πολλά, πολλά που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη, πρέπει να κάνουν αυτό που είναι στο καθήκον τους, όπως μιλείς, ισχύει για την προστασία της εσωτερικής αγοράς, της παραποίησης προϊόντων κλπ. Μπορούμε να εποπτεύουμε γενικά, θεσπίζουμε προδιαγραφέ κλπ. Έχουμε και το EU Pilot, το σύστημα για να δούμε αν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία IPPC. Το είπε και, ο κ. Ζεϊβελίνη. Ήδη έφτασε ή καταφτάνει η, απάντηση σε μια δική σας ερώτηση που υπεγράφει με τον ε, κύριο Σιλβέστης Βαλτάσαρ και την κυρία Ματέρα και αν δεν έφτασε ακόμα θα φτάσει σε λίγα λεπτά αυτή η απάντηση όπου δίνονται σαφεί απαντήσει στο τι πρέπει να κάνει η Ιταλία, δηλαδή να εγγυηθεί την πλήρη και σωστή εφαρμογή τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην επικράτειά της, στι οδηγίε του 2008 όσον αφορά την πρόληψη και την ολοκληρωμένη μείωση τη ε, Έχουμε μέσα, όπω σα έλεγα, ελέγχου και επαλήθευση, θα το διάβασα έτσι σύντομα. Ε, θα φτάσει η πλήρη απάντηση, αλλά λίγο πολύ αυτό λέει ο συνάδελφός μου, ο κ. Ποτότσνικ, απαντώντας στις ερωτήσεις σας. Πάντα τώρα όσον αφορά τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της Ιταλικής κυβερνήσεως, απαντώντας τον ε, κύριο Γιάρ, ήδη εξετάζει την αδειοδότηση την περιβαλλοντική, η διαδικασία πράγματι είναι περιπλοκότατη η απλούστευση είναι η απάντηση για να μειωθεί ο χρόνο απαιτούμενο και διαδικασίε. Συμφωνώ λοιπόν με τι εκκλήσει σα, αλλά επαναλαμβάνω ότι χθε μίλησα επί μακρόν, συζήτησα με τον Υπουργό Περιβάλλον Ιταλία που μου βεβαίωσε αυτή τη θέση και απαντώ αφού μίλησα μαζί του. Δεν ε, βασίζομαι επί υποθέσεων, μίλησα μαζί του. Απαντώντα τώρα στον κύριο Μποστινάρου, πέρα από το πρόβλημα τη βιομηχανική πολιτική, στο σύνολό της, υπάρχει ένα θέμα που θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο έθεσε και η κυρία Σαρτόρη του level playing field των σωτήμων όρων ε, για τους ανταγωνιστές και του χάλιβα που εισάγουμε. Ε, από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο θα πρέπει οι εισαγωγείς να κοινοποιούν στα κράτη-μέλη πόσος χάλιβας έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες και αυτό βάσει ενός κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ελήξει τη 31 Δεκεμβρίου. Η ανανέωση δεν έχει αποφασιστεί ακόμα προσωπικά. Ε, είμαι υπέρ. Ε, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο και ο Επίτροπος ο κ. Ντεχούκτ που είναι υπεύθυνο για αυτό το θέμα θα μιλήσει γι' αυτό. Αν η πρόεδρος η κυρία Ματσόνη θέλει στο τέλος της συζητήσεως να στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία σύνοψη εκφράζοντας τις θέσεις της Επιτροπής Αναφορών από αυτού του θέματος, όπως έκανε η κυρία Σαρτόρη, αυτό θα είναι κάτι που θα μπορέσει να αξιολογηθεί και να μελετηθεί με τη, μετά τις δεούσεις προσοχής. Όσον αφορά ένα άλλο ερώτημα που ετέθη από την κυρία Ματέρα και τον κύριο Ριβελίνο στον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, για την Παγκοσμιοποίηση. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, πιστεύω ότι αυτό το ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι δεν αφορά ενδεχόμενη μείωση παραγωγικότητας της ήλβα, Δεν είναι θέμα από βιομηχανοποίησης, αλλά μία κρίση που δημιουργήθηκε από δομικά διαστατικά προβλήματα ή από αθέμητο ανταγωνισμό. Εδώ μιλάμε για μη σεβασμό των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Όπως ήδη είπα επί τη ευκαιρία της διαθεσμικής συνόδου κορυφής στον Μπάρι, όπου ο πρόεδρος της περιοχής και ο Υπουργός Βίνη και ο Υφυπουργός Βιτσέντη και τα συνδικάτα ε, και στο ΙΛΒΑ υπάρχουν άλλα προγράμματα, άλλα μέσα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όπως τα περιφερειακά ταμεία της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ε, όπως το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ήδη χρησιμοποιείται, και το Horizon 2020, όπου εκεί υπάρχουν ε, πόροι για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την έρευνα σε αυτό το τομέα. Έχω υπόψη επίσης και το ταμείο για το χάλιβα και τον άνθρακα, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Ήλβα μας είπε ότι προτίθεται να συμμετάσχει σε κάποια από αυτά τα προγράμματα και απομένει να δούμε τι θα κάνει. κ. Τζανόνι και εκείνος ε, έθεσε το ζήτημα του σεβασμού των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν το περίμενε τις δικαστικές αρχές. Το είπα και στην παρέμβασή μου αυτό και πρέπει να το επαναλάβω όλα αυτά που μπορούν να γίνουν συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Επιτροπή Αναφορών επανειλημμένα ε, ε, στράφει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται. Σήμερα ήρθε ο αντιπρόεδρο της να μιλήσει, διότι θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως η Επιτροπή πάντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε. Ε, ξεκίνησε η δικασία, λοιπόν αυτή της παράβασης και μετά ε, απόφαση του δικαστηρίου. Παρακολουθεί η Ευρώπη, βλέπει τι γίνεται. Και αν σήμερα η Ιταλική κυβέρνηση ε, προσαρμόζεται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, το έκανε διότι εκλήθη να συμμορφωθεί η Ιταλία. Όσον αφορά τους κανόνες για την προστασία της υγείας, επ' αυτού είναι κάτι που εργαζόμεθα άοκνα, όπως είναι ο κανονισμός REACH ε, που πολλές προσπάθειες μας υποχρέωσε να κάνουμε και υποχρέωσε τι επιχειρήσει να κάνουν πολλέ προσπάθειε. Είναι όμω ένα μέσο που όχι μόνο εγγυάται την ανταγωνιστικότητα, αλλά είναι ένα μέσο που εγγυάται και την προστασία τη υγεία των πολιτών μα. Όλε οι δράσει, όλη η νομοθεσία μα κατά τη παραποίηση και για τον έλεγχο τη εσωτερική αγορά για άλλα τα προϊόντα που προέρχονται εκτός Ευρωπα... από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησα και μια εκστρατεία. Περιοδικά ξεκινά μάλλον την τελευταία την ξεκίνησα αρχές Αυγούστου φέτος όσον αφορά την παραποίηση. Πριν ξεκινήσουν οι διακοπές και ε, έδειξα δύο παπούτσια που είχαν παραχθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αρκούσε να μυρίσει κανείς αυτά τα παπούτσια για να καταλάβει πόσο ξεπερνούσαν τα μέγιστα όρια των επιτροπωμένων καρκινογόνων σιών. Δέκα φορές ξεπερνούσαν τα όρια. Πρέπει να πω ότι όσον αφορά τις στοιχές, τις κανονιστικές, κάνουμε πολλά. Όμως ε, δεν υπάρχει αστυνομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν υπάρχει η οικονομική υπηρεσία αστυνομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δεν υπάρχει χωροφυλακή. Δεν έχουμε μέσα αστυνόμευση για να μπορέσουμε να κάνουμε εξακριβώσει. Θα πρέπει αυτό να το αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Εμεί μπορούμε και θα πρέπει να θεσπίζουμε καλέ προδιαγραφέ για την προστασία τη υγεία των πολιτών Θεωρώ ότι ο Επίτροπος ο κύριος Νταλής και η κυρία Στεστόρης Γκότζε, η Γενική Διευθύντρια, υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία με τη βιομηχανική πολιτική. Ζητήσαμε θυσίες να γίνουν από τη βιομηχανία μας. Θεωρώ ότι η ανταπόκριση ήταν θετική. Έχω για παράδειγμα πάντα το σύστημα REACH διότι είμαι υπεύθυνο άμεσα γι' αυτό και το επίπεδο του 20% που εν τη απουσία γενική συμφωνίας δεν μπορεί να αυξηθεί. Όμως αν υπήρχε γενική συμφωνία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε διότι εδώ πρέπει να είναι ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε αύξηση. Όμως πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα με τους κανόνες που έχουμε είναι εκείνα που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον στον κόσμο. Κανόνες ισορροπημένοι που χρησιμεύουν στο να αποφύγουμε και την ε, μετακίνηση των επιχειρήσεων, τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων εκτός Ευρώπης, που αυτό σημαίνει παρέμβαση υπέρ της αλλαγής του κλίματος. Εφόσον δεν υπάρχουν σύνορα για το κλίμα, αν οι μεγάλες βιομηχανίες πάνε να παράγουν γιατί φεύγουν από την Ευρώπη, πάνε να παράγουν αλλού, διότι είναι χρήσιμο ο χάλιβας, χρειάζεται και πολλά προϊόντα ε, και ακόμα και της ενεργοβόρου βιομηχανίας και εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακος και πάνε να παράγουν σε άλλα μέρη του κόσμου που δεν υπάρχουν οι κανόνες, σε αυτή την περιπτώση χάνουμε ε, ανταγωνιστικότητα και γίνονται τα πράγματα πολύ πιο χαλαρά όσον αφορά τη δράση κατά της αλλαγής του κλίματος. Χρειάζεται καλή ισορροπία, όπως υπενθύμιζε και η πρόεδρος Σαρτόρη και χαίρομαι που η Επιτροπή Βιομηχανίας ζητά μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την κατάσταση του Χάλιβα. Εάν υπάρχει συμφωνία, εγώ με τα χαράς να σας δείξω τι κάνουμε και να σας δείξω και τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που θα συζητήσει αύριο, όχι, μεθαύριο θα συζητήσει ε, το ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του Χάλιβα. Πιστεύω ότι απάντησα στα πάντα. Α, αν θέλετε μπορώ να σας πω ακόμα και τις λεπτομέρειες απάντησης του κ. Ριβελίνη. Ο κ. Ριβελίνη μάλλον ζητούσε τα χρήματα που έδωσε η Ιταλία, η Ιταλική κυβέρνηση. 336 εκατομμύρια για την από μόλις 187 για τη βελτίωση των υποδομών του λιμανιού, 30 για την μηχανική ε, αποκατάσταση και 119 για τις δραστηριότητε αποκατάστασης. Δεν είμαι σίγουρος αν έφτασε ήδη η κοινοποίηση αυτών των παρεμβάσεων, όμως θα χρειαστεί αυτά τα ποσά να ε, από αυτά τα ποσά Θα ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε και ο Επίτροπος Αλμούνια να δει αν οι κρατικές ενισχύσεις ε, ταιριάζουν ή όχι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πιστεύω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, όμως το γραφείο μου κυρία Πρόεδρα και η γενική μου διεύθυνση είναι πάντα στη διάθεσή σας, στη διάθεση επιτροπής σας, την επιτροπή της οποίας προεδρεύετε για να δίδουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και όλες τις υποθέσεις που θα θεωρήσετε σκόπιμο να επιστήσετε την προσοχή μου επ' αυτών, της Γενικής Διεύθυνσής μου και του Γραφείου μου. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου, οι Επίτροποι, ε, είναι εξίσου διαθέσιμοι να συνομιλήσουν με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ εκ νέου που με επιτρέψατε να επιστρέψω και να συναντηθώ σε μια επιτροπή στην οποία ανήκα επί μια πενταετία. Είναι πάντα χαρά για μένα ε, να επιστρέφω στον τόπο αυτό που είχα εργαστεί υπέρ των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Αντιπρόεδρε, λέει η Πρόεδρο, πολύ συχνά λοιπόν θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη χαρά σα και θα σα καλέσουμε και άλλε φορέ να συμμετάσχετε στι εργασίε μα, δίνοντά σα την ευκαιρία να ξαναζείτε τι εμπειρίε του παρελθόντο. Μην κάνετε να ζηλεύει η πρόεδρο ε, Σαρτόρη, που έρχομαι πιο πολύ στη δική επιτροπή από ότι στην Επιτροπή Βιομηχανία. Για μας είναι χαρά, λέει η κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρέμβαση, για την υπόθεση Ήλβα και για το θέμα της κρίσης στον τομέα του Χάλιβα που περνάει η Ευρώπη, για τις απαντήσεις που μας δώσατε, για τη δεσιμότητά σας και για, σε μελλοντικέ ε, ευκαιρίε που υπάρξουν για να εκμεταλλευτούμε αυτά που θα μας πείτε, όπως μας είπατε σήμερα. Η συζήτηση για την αναφορά μπορούμε να την κλείσουμε Δεχόμενη μόνο την πρόταση του Αντιπροέδρου του κυρίου Ταγιάννη, που θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να υποστηρίξουμε, να παρουσιάσουμε και εμείς σαν Επιτροπή ε, μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου θα ζητούμε ε, βάσει τις συζητήσεις που έγινε σήμερα μια παρέμβαση πιο στοχευμένη και από την άλλη πλευρά την πρόταση για ένα ψήφισμα στην Ολομέλεια που θα μπορούσε να διατυπωθεί, να συνταχθεί την Επιτροπή μας και θα μπορούσε ίσως ε, να συζητηθεί από κοινού με την Επιτροπή ΕΝΒΗ τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να υποβάλουμε στην Ολομέλεια το ερώτημα που η Πρόεδρος ε, Σαρτόρη μας ανακοίνωσε, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε στην Ολομέλεια του ε, Στασβούργο να έχουμε μια συζήτηση επικεντρώνεται επί του τομέα του Χάλιβα, όχι μόνο για να καθορίσουμε μια νέα στρατηγική βιομηχανική, αλλά και για να συνδυάσουμε τη βιομηχανική πολιτική με τον πλήρη σεβασμό των αρχών για την προστασία της υγείας, της ζωής και του περιβάλλοντος ε, που είναι στο επίκεντρο του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρχουν αντίρρησεις, μπορούμε να κλείσουμε με αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ όλους Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Γκιωταγιάννη. Γεια σας.